Ε, Καλημέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά. Διότι έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό καλεσμένο και καλό θα ήταν να μην τον κάνουμε να περιμένει τόση ώρα. Όπως γνωρίζετε το Μαρόκο από το Μάρτιο ξεκίνησε μια διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης η οποία εξελίσσεται με την Επιτροπή Διαβούλευσης είναι συμβουλευτικό όργανο, συμμετέχουν γενικά πολιτικές οργανώσεις, οργανώσεις της νεολαίας, επιστημονικοί σύλλογοι, όμιλοι, και κατέθεσε ένα σχέδιο αναθεώρησης το οποίο υιοθέτησε ο Βασιλεύς και στις 10 Ιουνίου μετέφερε το έγγραφο αυτό στην κοινή γνώμη και στις αρμόδιες, στα αρμόδια όργανα δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο, παραμένει ε, φυσικά ο Άναξ αρχηγός του κράτους, αρχηγός του στρατού και επίσης αρχηγός της πίστης, θρησκευτικός ηγέτης δηλαδή. Παρ' όλα αυτά εισάγει και πολλά επιπλέον στοιχεία όπως η ανεξαρτησία του δικαστικού, ο διαχωρισμός του εκτελεστικού, του νομοθετικού και του δικαστικού σώματος και εισάγει επίσης ένα καθοριστικό θα έλεγα στοιχείο το οποίο θα οδηγήσει στη γυτνίαση του μαροκινού συστήματος το δικό μας στο σύστημα ισότητας ανδρών γυναικών. Στην ομιλία την οποία έκανε η αυτού μεγαλειώτη την προηγούμενη Παρασκευή ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό και όπως είπε, θεωρεί ότι είναι τα θεμέλια για μια συνταγματική, δημοκρατική, κοινοβουλευτική και κοινωνική μοναρχία. Υπογράμμισε το θέμα της, του διαχωρισμού των εξουσιών και της ισορροπίας των εξουσιών απαραίτητων για την δημοκρατική λειτουργία και προέβλεψε και ένα δημοψήφισμα τον επόμενο Ιούλιο. Αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, αλλά το κίνημα της 20ης Φεβρουαρίου θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές, έτσι όπως προτείνονται, δεν είναι επαρκείς και την επόμενη Κυριακή οργανώνεται μια διαδήλωση εναντίον του σχεδίου συντάγματος. Σε αυτά τα πλαίσια μας τιμά η παρουσία μιας αντιπροσωπείας από το Μαρόκο, της οποίας ηγείται ο Ντρίς Λαλαγκάρ και ο οποίος συνοδεύεται από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών, την οποία ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε. Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο αυτό προβλέπει νέες αρμοδιότητες για το Κοινοβούλιο, δικαίωμα πρωτοβουλίας για αναθεώρηση του συντάγματος, δικαίωμα να χορηγεί αμνηστία και επίσης να δημιουργεί, να ιδρύει επιτροπές έρευνας. Όλα αυτά είναι σημαντικά, θέλουμε τα σχόλιά σας πάνω στο σχέδιο αυτό και θα θέλαμε να μάθουμε ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα προκαλέσει το Σύνταγμα αυτό στην κοινωνία του Μαρόκου και στα πλαίσια των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ με την, για την ομιλία σας, θα την ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακαλώ μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά αν μπορείτε, γιατί θα υπάρχει και διαδοχική μετάφραση, βέβαια θα είμαστε λίγο ελαστικοί στον σεβασμό του χρόνου της ομιλίας σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντζάρη για την ε, την πρόσκλησή του. Ευχαριστούμε επίσης τους ε, βουλευτές ε, και τον πρόεδρο. أن أكون أمام هذه اللجنة المحترمة لأنه سبق لي أن حضرت منذ أربع سنوات أمام هذه اللجنة J'ai de nouveau l'honneur de euh, venir intervenir au... Θέλω να παρέμβω στην Επιτροπή αυτή διότι έχω συμμετάσχει ήδη πριν από τέσσερα χρόνια σε μία συνάντηση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τότε ε, υπήρχε <clears throat> μία περίοδος μεταβάσεως προς την δημοκρατία ε, σε όλη την Μεσόγειο και επιπλέον υπήρχε ένας εκπρόσωπος της Αλγερίας, της Τινησίας και ένας εκπρόσωπος της Παλαιστίνης πέραν ημών. Τώρα μετά από τέσσερα χρόνια από όταν ξεκίνησε η περίοδος ε, μεταβάσεως προς την δημοκρατία έχουμε επιτύχει μία σημαντική πρόοδο και επιπλέον όσον αφορά το θέμα των γυναικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η χώρα μας επιπλέον ε, προέβη σε μεταρρυθμίσεις οικονομικές και κοινωνικές που είναι πολύ σημαντικές και έχετε υπάρξει ένας στρατηγικός εταίρος πολύ σημαντικός για εμάς. Σήμερα λοιπόν προσχωρούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ε, σαν εταίρος επί του θέματος της δημοκρατίας. Ο αραβικός κόσμος αντιμετωπίζει ακόμη ορισμένα κινήματα αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στον αραβικό κόσμο συνέβη πριν μία δεκαετία στο Μαρόκο. Και εάν στον αραβικό κόσμο υπάρχουν ε, εβδομαδιές ε, ε, εκδηλώσεις και διαδηλώσεις. Αυτό συνέβη καθημερινά προδεκαετία στο Μαρόκο. Και από την ανεξαρτησία της η χώρα αντιμετωπίζει την εξής διαμάχη. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πίστευαν ότι έπρεπε καταρχήν να καταρτιστεί το κράτος, δηλαδή η διοίκηση και ο στρατός. Και επιπλέον αυτοί οι οποίοι από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι κάθε κατάρτιση κράτους περνά από την δημοκρατία. Και αυτό διαπιστώνεται μέσω μιας σημαντικής διενέξεως που κατέληξε σε σημαντικές συνέπειες, συλλήψεις και μία κατάσταση την οποία το Μαρόκο χαρακτηρίζει σαν χάλκινα χρόνια. και ε, αυτό το ξεπεράσαμε και ε, περίοδο περίοδο πολύ δυσάρεστη διότι στον αραβικό κόσμο αυτές ε, οι, οι ε, κινήσεις ε, ε, οδήγησαν σε έξαρση της αντιπολιτεύσεως ενώ εμείς πάντοτε ε, προωθούσαμε την ποικιλομορφία και στα πλαίσια αυτά έγινε 9 Μαρτίου και η ομιλία την οποία απίφθινε η αυτού μεγαλειώτης ο Βασιλέας και άνοιξε το δρόμο ε, για μια εθνική ε, συζήτηση υψηλού επίπεδου με ε, όλα τα πολιτικά κόμματα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των, της κοινωνίας των πολιτών. Στο τέλος αυτού του διαλόγου ε, υπήρξε η κατάρτιση του νέου ε, σύνταγμα το οποίο ανακοίνωσε ο βασιλέας στις 19 Ιουνίου. Οι μεγάλοι άξονες ε, του, του, της μεταρρύθμισης αυτής είναι η εξής. Πρόκειται ε, για ένα σύνταγμα το οποίο αποβλέπει στην αναμόρφωση του κράτους για μία νέα ανακατανομή των εξουσιών και εφαρμόζει τις βασικές αρχές του κράτους αναγνωρίζοντας την ε, ποικιλομορφία ε, των ταυτοτήτων του Μαρόκου Αραβική, ε, Βερβέρων, Χασεμίτων και Εβραίων. Και ε, από την Ανδαλουσία και Μεσογειακή. είναι η αναγνώριση της ε, γλώσσας των Βερβέρων σαν δεύτερη επίσημη γλώσσα του κράτους πέραν των Αραβικών και ε, πρόκειται ε, για ένα πραγματικό χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη και που ενισχύει την ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, αναβαθμίζοντας την ε, ισότητα των φύλων και η εθνική κυριαρχία όπου προέχει το Σύνταγμα που διατυπώθη μέσω του δημοψηφίσματος και των ελευθέρων εκλογών όπου προέχει το Σύνταγμα επί όλων των αρχών και όλων των θεσμικών οργάνων όπου υπάρχει μία, ένας διαχωρισμός των εξουσιών μεταξύ της κοινωνικής και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και στα πλαίσια αυτά υπάρχει μία κατάργηση όλο, κάθε αναφοράς στον ιερό χαρακτήρα του, του ατόμου του βασιλέα και ε, ε, διαχωρισμό των ε, θρησκευτικών εξουσιών. Η νομοθεσία λοιπόν παρέμεινε αρμοδιότης απλώς του Κοινοβουλίου και μοναδικά. Η κυβέρνηση προέρχεται από ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο και ο αρχηγός της ε, κυβέρνησης ε, ε, καθορίζεται από το Κοινοβούλιο και από το κόμμα το οποίο υπερίσχυσε στις εκλογές με πλήρεις εξουσίες εκτελεστικές. Πρέπει λοιπόν να κατατιστεί μια γενική πολιτική και να υπάρχει επίβλεψη όλων των διοικητικών θεσμικών οργάνων. Χρειάζεται ένα ισχυρό κοινοβούλιο με ενισχυμένες εξουσίες που θα εξασκεί όχι μόνο το νομοθετικό έργο αλλά θα ελέγχει το, η κυβέρνηση και θα αξιολογεί ε, τις ε, δημόσιες πολιτικές. που θα, θα ενισχύουμε ε, την αντιπολίτευση, θα ενισχύσουμε και το ρόλο της αντιπολιτεύσεως στο Κοινοβούλιο και η ε, δικαιοσύνη έχει επίσης καταστεί ε, εξουσία για να εξασφαλίζει την διαφύλιξη των δικαιωμάτων και του νόμου. Εξού και υπήρξε μία πλήρης, ένας πλήρης διαχωρισμός των εξουσιών των δικαστών. Ε, περαιτέρω δημιουργήθηκε ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο θα παρακολουθεί την, και θα αναλάβει την προστασία ε, του συντάγματος και της εφαρμογής του. Αυτό το οποίο είναι νέο στοιχείο σε αυτό το σχέδιο συντάγματος είναι η συμμετοχική δημοκρατία. και ε, δίδεται στα πλαίσια αυτά η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις για νομοσχέδια και για κατάρτιση νόμων και αναγνωρίζεται δηλαδή μέσω του νέου συντάγματος η σημασία της κοινωνίας των πολιτών, ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων Ε, υιοθετείται η αναγνώριση του ρόλου των μέσων ενημέρωσης στην ε, προστασία των ελευθεριών των ε, πολιτών και δημιουργείται ένας νέος τομέα συμμετοχικής δημοκρατίας για την παιδεία, την κοινωνία και την νεολαία και ε, επιπλέον ε, ε, κατανέμεται σε περιφερειακό επίπεδο κατανέμονται ορισμένε αρχές και είμαστε καταρχήν στον τομέα της χρηστής διακυβέρνησης. Όλα αυτά χωρίς ε, να καταρρεύσει η συνταγματική βασιλεία σαν πολίτευμα η οποία εξασφαλίζει τις πολιτικές ε, μεταρρυθμίσεις αναφέρεται στην νομοθεσία για τις πολιτικές ομάδες, για τον εκλογικό νόμο, για τα μέσα ενημέρωσης και όλοι, όλοι αυτοί οι νόμοι που περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο συντάγματος αποτελούν 26 νέους οργανικούς νόμους και αυτοί οι νόμοι θα θα προβούν εις ε, την ε, πολιτική μεταρρύθμιση, θα εξασφαλίσουν την πολιτική μεταρρύθμιση. الوطني للأحرار الأستاذ حسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية دريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المجتمع المدني. Encore une fois, merci beaucoup et. Euh... Και με αυτά ολοκληρώνω την ομιλία μου και ε, θα είμαστε στη διάθεσή σας ολόκληρη αντιπροσωπεία να απαντήσει στις ερωτήσεις σας μαζί με τον ε, Γενικό Γραμματέα ε, του Εθνικού Κόμματος Ανεξαρτήτων και το εκπροσώπου ε, του Συνταγματικού Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Ξεκινάμε με τον κύριο Σαλαφράνκα, συντονιστή του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών και σας καλωσορίζω. Θα ήθελα να κάνω γενικά μια ερώτηση. Ε, πώς αξιολογείτε τη ε, μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή, μεγαλύτερη δημοκρατία. Ε, εσείς γνωρίζετε την ε, μεσογειακή πολιτική, τη νέα πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόσφατα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Πώς σας φαίνεται αυτό. Ε, στη συνέχεια σημειώνουμε με ενδιαφέρον ε, τη συνταγματική μεταρρύθμιση που θα ψηφιστεί την 1η Ιουλίου. Όπως είπατε, ο Βασιλεύ δεν θα είναι ε, ιερό πρόσωπο, απλώς απαραβίαστο. Απλώς θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημασία αξίζει να δώσετε ε, τα γεγονότα που συμβαίνουν στις γειτονικές σας χώρες. Μας είπατε ότι είχατε έρθει ε, συνοδευόμενος από ε, εκπροσώπους των γειτονικών χωρών σας και ε, Παλαιστίνιους. Αυτά που συμβαίνουν στην Τινησία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, πώς τα αξιολογείτε και σε άλλες χώρες και πώς μπορούν αυτά να επηρεάσουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Αραβικού Μαγρέμπ. Ε, Στο άρθρο 41 ε, του σχεδίου συντάγματος διασφαλίζεται η ανεξιθρησκεία και η ελευθερία. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, το άρθρο αυτό και στο πνεύμα ή στο γράμμα του επίσης εγγυάται ε, τη δυνατότητα ελευθερία συνείδησης, δηλαδή να μπορεί κάποιος να αλλαξοπιστήσει. Και επίσης ποια είναι τα κινήματα εκείνα που στο εσωτερικό της χώρας σας αντιτίθεται σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Βεβαίως το κίνημα των νέων της 20ης Φεβρουαρίου η δημοκρατική οδός, ένα άλλο κείμενο και ένα τρίτο και τελειώνω Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Υπουργέ κάτι για το άρθρο 90 του εκλογικού κώδικα. Επιτρέπει κανείς να κάνει προεκλογική εκστρατεία κατά της μεταρρύθμισης του συντάγματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε αρκετό χρόνο για να δώσουμε την, τον λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Να προσθέσω εδώ ότι ανάλογα με το τι επιθυμείτε κύριε Υπουργέ, μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις και τα μέλη των αντιπροσωπιών σας, ίσως σε ειδικά θέματα, πάνω στα οποία έχουν συγκεκριμένες γνώσεις και αρμοδιότητες. Η κυρία Έιτς έχει το λόγο, η συγγήτριά μας για την συμμετοχή του Μαρόκου στα κοινοτικά προγράμματα και συντονίστρια της φιλελεύθερης ομάδας. Κυρία Νέιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μέλη της Αντιπροσωπείας, να σας καλωσορίσω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω επίσης ξεκινώντας την ικανοποίησή μου, να αναφερθώ στην ικανοποίησή μου μετά την ανάγνωση της ομιλίας της αυτού μεγαλειότητας και των προτάσεων των μεταρρυθμιστικών τις οποίες περιλαμβάνει. Όπως γνωρίζει ο κύριος Πρέσβης, το Μαρόκο είναι μια χώρα που εγώ και ο σύζυγός μου γνωρίζουμε πολύ καλά. Την επισκεφτήκαμε για πρώτη φορά πριν από 40 χρόνια. Είδαμε τη χώρα σας να αλλάζει προς την καλύτερη συνήθως κατεύθυνση και αυτό το σχέδιο συντάγματος και οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται είναι προτάσεις τις οποίες κάποιες άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες δεν μπορούν καν να ονειρευθούν. Βρίσκω λοιπόν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες τις ε, προόδους τις οποίες επιτελεί το πρόγραμμα. Βέβαια δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων, ιδιαίτερα των ηγετών του κινήματος της 20 Φεβρουαρίου, αλλά σαφώς και υπερβαίνει κάποια, τα οποία, κάποια όρια τα οποία εμείς αναμέναμε να ισχύσουν. Υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες βέβαια εδώ και θα ήθελα να σας θέσω γι' αυτό κάποιες ερωτήσεις. Το πιο σημαντικά θα πρέπει να ακολουθήσουν η εφαρμογή δηλαδή όλων αυτών των προτάσεων. Ένα παράδειγμα να δώσω. Στο σχέδιο συντάγματος προβλέπεται ότι θα απαγορεύεται στους βουλευτές να αλλάζουν κόμμα κατά τη διάρκεια της νομοθετικής περίοδου εντολής. Πρόκειται για μια σημαντική θα έλεγα περιοριστική ε, ρύθμιση λόγω των εξελίξεων των πολιτικών τα τελευταία πέντε χρόνια βλέπουμε να δημιουργούνται νέα κόμματα. Κόμματα τα οποία φυσικά δημιουργήθηκαν και με την, ε, ελπίζω να μην ε, θίξω κανέναν, αλλά με πρόσφυγες πολιτικούς που ήρθαν από άλλα κόμματα. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν στην περίπτωσή σας. Έχει σημασία λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι Μαροκινοί, παρουσιάζεται παντού και στη δική μου χώρα και στη δική σας φυσικά κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί μια τέτοια διάταξη. Δεύτερον, για να διασφαλιστεί η διάρκεια της δημοκρατίας στο Μαρόκο θα είναι θεμελιώδες τα διαφορετικά πολιτικά κόμματα, τα διάφορα συγγνώμη πολιτικά κόμματα, θα είμαι πολύ ειλικρινής εδώ, να κάνουν περισσότερες προσπάθειες από όσες έκαναν μέχρι τώρα έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τους Μαροκινούς και των δύο φίλων και της πόλης και των χωριών της Υπέθρου να εγγραφούν ως ε, ε εκλογής και να συμμετέχουν στις εκλογές. Ε, το πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές είναι κάτι το οποίο τίνει στο να εξασθενήσει θα έλεγα την ε, διασφάλιση της διάρκειας ε, της μαροκινής δημοκρατίας. Και ένα τελευταίο στοιχείο και τελευταία ανησυχία, το πρόγραμμα προωθεί την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του τύπου. Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίσαμε ε, κάποιες ειδήσει ε, εις βάρος δημοσιογράφων, δίκες εις βάρος δημοσιογράφων, δίκες και διώξεις εις βάρον αρχισυντακτών περιοδικών. Αυτά είναι λίγο αντιφατικά μεταξύ τους. Πώς τα σχολιάζετε παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Νέιτς. Ο κύριος Γιάννες, πρόεδρος της διάσκεψης των προέδρων των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ και όλη την αντιπροσωπεία από το Μαρόκο που είχε τη γαλοσύνη να έρθει ε, και να παραστεί στη σημερινή συζήτηση. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι Ισπανός και συγκεκριμένα από την Ανδαλουσία και αισθάνομαι πολύ κοντά μου το Μαρόκο, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και πολιτιστικά και γενικότερα και ε, έτσι συναισθηματικά. Θεωρώ ότι γνωρίζω αρκετά καλά το Μαρόκο και ό,τι συμβαίνει εκεί ε, το αισθάνομαι πάρα πολύ δικό μου και πάρα πολύ κοντινό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι λοιπόν και πολύ χαρούμενοι που είδαμε να αρχίζει αυτή τη διαδικασία συνταγματικής και πολιτικής μεταρρύθμισης ο βασιλεύς στη χώρα. Καθοδόν έτσι προς τη μετάβαση προς μια συνταγματική μοναρχία και κοινοβουλευτική μοναρχία. Οπότε θεωρώ ότι η χώρα βρένει προς σωστή κατεύθυνση και μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξή μας, στην συμπάθειά μας, στη στήριξη στο βαθμό που το χρειάζεται. Βεβαίω πρόκειται για ένα θέμα που αφορά κυρίως το μαρακινό λαό και ε, τους θεσμούς της χώρας. Κατόπιν τούτου, συμφωνώ και συνεχίζω από εκεί που ρώτησε η προλαλήσασα. Ένα ευαίσθητο σημείο σε κάθε δημοκρατία είναι η ελευθερία της έκφρασης και το θέμα της ελευθεροτυπίας και το Μαρόκο. Για να το πω έτσι, το έζησε ε, έτσι με τρόπο εύσχημο. Ε, το έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια και με δημοσιογράφους, με διευθυντές εφημερίδων και με εξόριστους δημοσιογράφους ε, που θέλησαν να αναφερθούν σε μια ευρύτερη μεταρρύθμιση. Και ένα άλλο πολύ ακαθόδες θέμα που γνωρίζω ότι ειδικά για το Μαρόκο είναι και ευαίσθητο και λεπτό και αυτό είναι η Δυτική Σαχάρα που θεωρεί το Μαρόκο δικό του έδαφος, δική του επικράτεια. Αλλά η διεθνή κοινότητα και οι Ηνωμένα Έθνη ε, θεωρούν ότι πρόκειται για μια επικράτεια, για ένα έδαφος όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η ε, αποχώρηση της απεικιοκρατίας. Γιατί μια δημοκρατία και πλήρης δημοκρατία δεν μπορεί να νοείται, ούτε μπορεί να συνίσταται χωρίς... Ε, να ε, έχει επιτευχθεί πρόοδο σε αυτό το ευαίσθητο και ακαθόδε θέμα. Αυτά, Υπουργέ, και σας ευχαριστώ και σας εγχαίρω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρέσβη, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την παρουσίαση την οποία κάνατε και να χαιρετήσω επίσης και την παρουσίαση από τον Μωάμεθ τον Έκτο του σχεδίου συντάγματος. Ξέρω ότι ήταν αναμενόμενο το σχέδιο συντάγματος. Πολλοί συνάδελφοι που συμμετέχουν στην διακοινοβουλευτική με το Μαρόκο ήμασταν ε, εκεί και είδαμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και όχι μόνο στο εσωτερικό του Μαρόκου αλλά και εκτός. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, μια μορφή εκδημοκρατισμού η οποία είχε, την οποία είχατε υποσχεθεί προς τον λαό της χώρας σας και πριν από την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ειρηνικής που θα οδηγήσει σε αλλαγές. Η απόδειξη αυτής της διαδικασίας είναι κάτι το πολύ θετικό για όλους και για μας. Και έτσι μπορούμε να κρίνουμε και με συγκριτικό τρόπο αν θέλετε τις διάφορες αλλαγές στην περιοχή και στον αραβικό κόσμο ευρύτερα. Δεν μπορώ φυσικά να κάνω μια πλήρη αξιολόγηση όλων των αλλαγών οι οποίες προτείνονται. Πρόκειται για ένα σύνταγμα το οποίο γίνεται πολύ πιο σύνθετο, 180 άρθρα σε σχέση με τα 68 τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα. Ε, θεωρώ όμως 148 euh, είναι μάλλον τα άρθρα του συντάγματος από 68 που ήταν. Πάντως ε, δημιουργείται ένα σύστημα ίδιων του Μαρόκου και των ειδικών του χαρακτηριστικών. Και υπάρχει επίσης και αναφορά ε, για την καλύτερη συνεργασία και στενότερη συνεργασία με τις χώρες στα πλαίσια της ε, τις γειτονικές χώρες και την ευρύτερη περιφέρεια. Αυτό λοιπόν είναι για πρώτη φορά ίσως περιλαμβάνεται στο συνταγματικό πλαίσιο μιας χώρας και αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές του Μαρόκου και προς την Ευρώπη είναι πολύ συγκεκριμένες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα πολύ θετικό μήνυμα και να υπογραμμίσω ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεσμοποιείται θα έλεγα Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς μας στη χώρα σας συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου του Εθνικού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και νομίζω πως το ότι το όργανο αυτό υποστηρίζεται πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν μέσω αυτής της θεσμοποίησης είναι κάτι το πολύ θετικό και αυτά τα οποία προβλέπονται για την ισότητα των φύλων και η δημιουργία μιας επιτροπής ισότητας είναι και αυτά πολύ θετικά βήματα. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε μια συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει σχετικά με το προφίλ αυτού του καθεστώτος. Κάποιοι λέγουν ότι έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο παραπέμπει στην πέμπτη προεδρική γαλλική δημοκρατία χωρίς τις εκλογές ανά πενταετία. Άλλοι πιστεύουν ότι δεν έχει καμία σχέση, υπάρχουν οι ασκούν κριτικοί και οι οποίοι θα ήθελαν να καταργηθεί πλήρως ο πολιτικός ρόλος της Βασιλείας. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια πιο ξεκάθαρη αντίληψη για τον διαχωρισμό των εξουσιών και να χαιρετήσω επίσης εδώ και την δημιουργία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες παρουσιάζονται για τη διασφάλιση της ελευθερίας της δικαστικής εξουσίας. Ε, συνεργάστηκα με τον συνάδελφο Αμπτεραχμάν Αχμούντ σχετικά με την αποκέντρωση η οποία θεσμοποιείται σε επίπεδο ε, εθνικό και ξέρουμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στη Να κάνω τρεις σύντομες παρατηρήσεις εδώ, μικρές ερωτήσεις ίσως, τις οποίες θα μου επιτρέψετε να σας απευθύνω. Το πρώτο αφορά την διαδικασία της συζήτησης, του διαλόγου. Ο βασιλεύς αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει διάλογος. Υπάρχει μια χρονική περίοδος πριν από το δημοψήφισμα λοιπόν και δεν ξέρω ακριβώς πώς θα οργανωθεί η συζήτηση αυτή σε σχέση εν πάση περιπτώσει με ε, το περιεχόμενο των προτάσεων. Μέχρι τώρα οι συζητήσεις γινόντουσαν σε ένα ακαθόριστο πλαίσιο. Τώρα πλέον ε, το πλαίσιο αυτό γίνεται πιο συγκεκριμένο. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα του ποσοστού συμμετοχής. Το ποσοστό συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά, χαμηλό. Ξέρετε αν τώρα μετά από αυτήν την παρέμβαση του βασιλέως θα αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής νομιμοποιεί θα έλεγα την διαδικασία του δημοψηφίσματος. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν θα περάσει ή όχι το δημοψήφισμα, ο λαός καταφατικά θα απαντήσει στις ερωτήσεις, αλλά το θέμα είναι το ποσοστό. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους αντιτιθέμενους. Ξέρουμε ότι το κίνημα της 20ης ε, ε, Φεβρουαρίου συνεχίζει, δεν έχει ηρεμήσει σε εισαγωγικά. Πώς εσείς θα προσπαθήσετε να συμπεριλάβετε στη διαδικασία που θα ακολουθήσετε το κίνημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Έχω μία ερώτηση η οποία βαίνει προς άλλη κατεύθυνση, η οποία όμως ε, εφόσον μου δίδεται σήμερα η ευκαιρία μου φαίνεται σημαντική. Με συγχωρείτε που άργησα να έρθω, αλλά συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο και στις επόμενες ημέρες πρέπει να διατυπώσουμε μία γνωμοδότηση για να δούμε αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνενέσει ή θα απορρίψει αυτή τη συμφωνία. Βλέπω ότι έχετε κάνει προόδους και αξιέπαινες και ε, που βαίνουν προς μία θετική αλλαγή. Το θέμα της Δυτικής Σαχάρα ήδη έχει αναφερθεί, ε, περιλαμβάνεται ε, εις ε, τις διαπραγματεύσεις για αυτήν την εμπορική συμφωνία, αλλά θα ήθελα να ξέρω και ρωτώ την γνώμη σας. Πιστεύετε ότι καλό θα ήταν να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε για αυτή τη συνεργασία γρήγορα ή θα ήταν καλύτερα για την ε, ε, αλλαγή της πολιτικής να πούμε ότι προτού προχωρήσουμε στο σημείο αυτό χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις διότι όντως υπάρχει μία πορεία προς μία πολύ θετική εξέλιξη και κατά αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι της χώρας θα υποφεληθούν της συμφωνίας όπως άλλωστε και η υπέρθρος η οποία θα μπορέσει να αποκομίσει μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σκόπιμο, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα σε τρεις πολύ σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες είναι παρούσες εδώ και αντιπροσωπεύουν μερικές φορές και μία διαφορετική άποψη από αυτήν της κυβέρνησης Πρόκειται για εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ξεκινήσω από τον Λασέν Νταουντή, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος του κόμματος της δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μοχάμεν Νταουτζάρ, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Ανεξαρτήτων. Παρακαλώ πέντε λεπτά ο καθένας, μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές και εκείνους που δεν μίλησαν. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια προς τη χώρα μου και για τη συμπάθεια και την αγάπη που μας έχετε βεβαιωθείτε ότι είναι αμοιβαία. δε μάλλον που ε, πολλοί Μαροκινοί σπούδασαν στην Ευρώπη. Μιλούν ευρωπαϊκές γλώσσες βλέπουμε ότι ε, έχουμε και καθολικό γάμο μεταξύ Μαρόκου και ε, Ευρώπης και κοινωνία γενικότερα. Λοιπόν, ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις που είναι και πολλές, αλλά να πω καταρχάς ότι όταν γίνεται λόγος για το Μαρακινό Σύνταγμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που ζείτε εσείς είναι πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς λέγουμε και τα θεωρείτε αυτονόητα. Δεν είναι για μας αυτονόητα όμως, γιατί πρόκειται για το Σύνταγμα του 1996. Το σημερινό Σύνταγμα είναι επανάσταση σε σχέση με το Σύνταγμα του 1996, διότι υπογράψαμε συμφωνίες για προεγμένη συνεργασία με την Ευρώπη και μάλιστα σήμερα ε, και έρχομαι από το Στρασβούργο ε, σήμερα, το Μαρόκο δεν έχει άλλη επιλογή παρά να προσεγγίσει την Ευρώπη. Υπογράψαμε λοιπόν Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και ε, πανψηφί στο Κοινοβούλιο, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα με την Ευρώπη. Ενώ ε, όταν πρόκειται για τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με τις Ηνωμένε Πολιτείε επί το κόμμα μου το καταψήφισε. Καταλαβαίνετε γιατί. Η Ευρώπη για μας λοιπόν είναι στρατηγικός εταίρος και το δικό μου κόμμα ε, της ε, δικαιοσύνης και της προόδου θεωρείται και Ισλαμιστικό κόμμα ε, και σας λέω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά, δεν θα χρησιμοποιήσω ξύλινη γλώσσα. Μ' αρέσουν όλες οι γλώσσες εκτός από την ξύλινη. Τι συμβαίνει στον αραβικό κόσμο και πώς αυτό επηρεάζει το Μαρόκο. Ο αντίκτυπος θα ήταν πραγματικά ολέθριος εάν δεν είχαμε αρχίσει αυτή τη διαδικασία εκδημοκρατισμού σε συνεργασία με την Ευρώπη. Γιατί και η Ευρώπη γνώρισε δικτατορίες. Ε, και τις βοήθησε. Η νησία δεν άξιζε τη βοήθεια, ούτε το Αιγυπτιακό καθεστώς. Ευτυχώς σε συνεργασία με την Ευρώπη τη γλίτωσε φτηνά το Μαρόκο. Και ε, θέλουμε να προχωρήσει ο εκδημοκρατισμός και θέλουμε το Μαρόκο να είναι μοντέλο, να είναι πρότυπο, να είναι η κινητήριος δύναμη. Είμαστε ο καλός μαθητής του αραβικού κόσμου ή της αραβικής τάξης. Βεβαίως δεν έχουμε το Ισπανικό Σύνταγμα, αλλά έλεγα προηγουμένως στους δημοσιογράφους ότι εμείς είμαστε η Ισπανία του αραβικού κόσμου. Έχουμε μια μοναρχία ε, ισπανικού τύπου στον αραβικό κόσμο. Προχωρούμε λοιπόν. Φανταστείτε ότι αρχίζει σιγά σιγά να διαχωρίζεται ε, η θρησκεία από το κοσμικό στοιχείο. Δεν υπάρχει φετφάς, δεν υπάρχει ε, δυνατότητα δυνατότητα ε, ερμηνείας ε, θρησκευτικών ε, γραφών παρά μόνο αμέσω του βασιλέως. Δηλαδή ο βασιλέας είναι κάτι σαν τον Πάπα, εκτός αν πείτε για το στρατό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να επεμβαίνει ο στρατός. Αυτό θα κατοχυρωθεί σε επόμενη αναθεώρηση. Έχουμε ένα πρωθυπουργό που είναι υπόλογος ενώπιον του λαού. Η κυβέρνηση δεν είναι πλέον υπόλογη στο βασιλιά, αλλά αποκλειστικά στο κοινοβούλιο. Για μας είναι μεγάλη αλλαγή αυτό. Θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο και θα έρθει και αυτό, θα γίνει. Είπαμε, δεν θέλουμε η χώρα να θεωρείται Ισλαμική χώρα, μουσουμανική χώρα. Ο, ο βασιλεύς είναι ο ηγέτης των πιστών. Δεν μπορεί να είναι κοσμική η χώρα μας, γιατί αλλιώς ο καθένας θα μπορεί να ερμηνεύει το Ισλάμ. Εμείς είπαμε αν είχαμε, αφήσει, αν είχαμε ζητήσει να αφαιθεί ελεύθερη ερμηνεία του Ισλάμ μπορεί να παίρναμε και 60% αλλά αυτό που θέλουμε είναι να παραμείνει στα χέρια του βασιλέως. Αλλιώς θα ε, είναι πολύ μεγάλη η ε, κούρσα των πολιτικών κομμάτων και για αυτό το θέμα. Και συμφώνησαν οι αρμόδιες αρχές στο Μαρόκο γιατί θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά, να προσεγγίσουμε την Ευρώπη αλλά να γίνουν όλα αυτά με κάποια πλαισίωση, με συνοδεία διότι η δημοκρατία είναι και οικονομική δημοκρατία. Διότι με την ένδυα καταλαβαίνετε ότι είναι πρόσφορο έδαφος αυτή για οποιαδήποτε ιδεολογία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στο Μαρόκο. Κυρία μου, μιλήσατε για τις συμφωνίες. Εγώ είμαι οικονομολόγος και θα μου επιτρέψετε με κάθε ταπεινότητα να πω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και τον αγροτικό κόσμο, γιατί έχουμε πλέον ένα πράσινο γεωργικό Μαρόκο, θα βοηθήσει τους αγρότες. Ξέρετε ότι είναι μικρή αγορά στο Μαρόκο, χρειαζόμαστε μια αγορά δίπλα μας. τώρα έχουμε εντάξει βιομηχανικές και οικονομικές συμφωνίες, θα επιθυμούσαμε και γεωργικές. Και θα επιθυμούσαμε οι Ισπανοί μας φίλοι να καταλάβουν ότι θα πρέπει και το Μαρόκο να μπει στο τρένο της Ευρώπης. Εγώ πήγα στην Ισπανία το 1971. Η Ισπανία συγχρονίστηκε. Ε, με την Ευρώπη. Κάποτε λέγαμε ότι η Ευρώπη είναι από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια. Ε, τώρα όμως, ε, αν θέλουμε μια Μεσόγειο ειρηνική, ε, θα πρέπει να βοηθηθούν και χώρες της Νότιας Όχθης Μεσογείου και προκειμένου το Μαρόκο και να μας υποστηρίζετε και να μας καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μοχάμεντα Ουτζάρ, Γενικός Γραμματέας του κόμματος της Εθνικής Ένωσης των Ανεξαρτήτων. Παρακαλώ μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξοχότατε. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε εφόσον ε, μας υποδεχθήκατε σε αυτή τη συνεδρίαση και ήρθαμε απλώς να σας μεταφέρουμε την ε, βαθιά πολιτική μας πεποίθηση ότι το Μαρόκο περνά από μια ιστορική περίοδο μεγάλης αλλαγής και μεγάλης εξελίξεως. Είχα την ε, τιμή ε, και την ευκαιρία να είμαι πολιτικά στρατευμένος υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της διαργασίας σαν εναλλακτικός πολιτικός και παρόλα τα αποτελέσματα, παρόλες τις προόδους ε, έχουμε μεγάλες, ε, δυνατο... Ε, μεγάλες δυσκολίες να πείσουμε τους νέους στο Μαρόκο να ακολουθήσουν και ε, να αφοσιωθούν ε, εις ε, την πολιτική αλλαγή. Οι νέοι δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι η πράξη της ψήφου διότι εφόσον όλα γινόντουσαν γιατί να ψηφίζει κανείς, γιατί να μετακινηθεί, γιατί να ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά η νέα μεταρρύθμιση αναρρύθμιση θα μας επιτρέψει να πείσουμε την νεολαία ότι, ότι ψηφίζοντας και συμμετέχοντας μπορεί κανείς ε, να επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές της χώρας και στον καθορισμό του Πρωθυπουργού. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να τονίσουμε τις ε, μεταφορές, τις μεταβιβάσεις ε, των ε, εξουσιών που, που θα μετατεθούν ή στον Πρωθυπουργό σαν αρχηγό της κυβέρνησης και έτσι οι νέοι θα μπορέσουν να λάβουν το μήνυμα, να αφοσιωθούν και να μεταφέρουν αυτή τη διδαχή στις διαδηλώσεις για να εκδιώξουν την διαφθορά και ε, να εφαρμόσουν μία πολιτική άξια αυτής της νέας νέας, της νεολαίας και γι' αυτό θέλω να χαιρετήσω το, την τόλμη του βασιλέα Μοχαμέτου Έκτου που κατάλαβε ε, τις ε, βλέψεις της νεολαίας. Όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα έχει το Μαρόκο τις καλύτερες ε, ε διαθέσεις για να μπορέσει ε, να ε, καταλήξει σε μία μία σχέση όπου θα υποφεληθούν και οι δύο πλευρές και θα λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των αλγερινών αδελφών μας και θα ε, δώσει μία σημαντική αυτονομία. Ε, έτσι θα υπάρξει ε, ένα προηγμένο πλαίσιο συνταγματικά που θα καλύψει εντός του συντάγματος το σχέδιο της αυτονομίας αυτονομίας της περιοχής. Συνεχίζουν οι συζητήσεις και δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε από τις άλλες πλευράς, από την πλευρά των Αλγερινών την ίδια πολιτική βούληση να τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία που είναι σημαντική. Και ε, που διεξάγεται υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών. Ή έχει έρθει η ε, Αραβική Άνοιξη, άρα και στο Μαγκρέμπ θα πρέπει να υπάρξει η Άνοιξη αυτή, η πρόοδος, η ελευθερία εκφράσεως και ελπίζω ότι από την άλλη πλευρά των συνόρων θα υπάρξει μια θετική αντίδραση και θα θα μπορέσουμε να έχουμε ε, μία δημοκρατική Αλγερία, ένα δημοκρατικό Μαρόκο και εξασφάλιση στο Μαγκρέμπ μίας αυτονομίας βάσει των αρχών που πρότεινε το Μαρόκο στα πλαίσια της κυριαρχίας του της εθνικής του κυριαρχίας. Ε, επίσης, ε, όντας στρατευμένος υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ελπίζω ότι θα υπερισχύσει το διεθνές δίκαιο και θα εφαρμοστεί στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο και στον κύριο Ντρίσελ Λιατζάμι, πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας. Θα ήθελα να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά τη συζήτηση γύρω από το Σύνταγμα και την προετοιμασία του δημοψηφίσματος. Υπήρξε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Υπουργών την Παρασκευή και αυτοί οι οποίοι ε, είναι κατά θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης πέραν της προσκλήσεώς τους σε συζητήσεις οι οποίες οργανώνονται από ιδιωτικά μέσα και δημόσια μέσα ενημέρωσης. Χθε αυτοί που πρεσβεύουν το όχι πήραν μέρος στο κρατικό κανάλι σε μια συζήτηση που κράτησε μια μισή ώρα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να διαφωτίσω και εγώ α, ε, τις απορίες σας σχετικά με το κίνημα της 20 Φεβρουαρίου. Κάποιοι από τους ηγέτες του κινήματος αυτού εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο συνταγματικό κείμενο να κάνω εδώ τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη. Εμείς θεωρούμε ότι η έκφραση διαφορετικής άποψης είναι απόδειξη πλουραλισμού. Θα ήταν σοβαρό σε ένα δημοκρατικό ε, σώμα να μην υπάρχει αντίθετη άποψη. Δεύτερον, θα ήθελα επίσης να θυμίσω, μιας και είμαι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής που οδήγησε στην σύνταξη του σχεδίου συντάγματος και που τροπολογήθηκε στη συνέχεια από τα πολιτικά κόμματα, να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η Επιτροπή αυτή <clears throat> έλαβε 185 μνημόνια. Αν πάρουμε τα 33 κόμματα και τα 5 συνδικάτα τα οποία έστειλαν μνημόνια, αυτό σημαίνει ότι 148 μνημόνια μας, προ... ήρθαν στα χέρια μας από την κοινωνία των πολιτών. Για να μπορέσει κανείς να καταλάβει καλά τη μαροκινή δυναμική θα πρέπει να την εγγράψει στα πλαίσια μιας πλουραλιστικής εικόνας, αλλά η κοινωνία των πολιτών, εκτός και αν παρανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί δεν ταυτίζεται με τους ηγέτες της 20 Φεβρουαρίου. Τώρα, είναι προφανές ότι εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να στηριχθεί η συνταγματική αλλαγή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Ποια είναι τα σημεία αυτά. Να θυμίσω ότι το σχέδιο του νέου συντάγματος ανοίγει με ξεκάθαρο τρόπο τις δυνατότητες συνταγματικής μεταρρύθμισης. Τα δύο σώματα δηλαδή από κοινού μπορούν συνεδριάζοντας να προχωρήσουν σε αλλαγές. Το θέμα είναι αν πράγματι θέλουμε να μπούμε σε μια πλουραλιστική και δημοκρατική λογική. Και μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με την ελευθερία συνείδησης. Πρέπει να το πούμε εδώ ξεκάθαρα. Το σχέδιο του νέου συντάγματος εγγυάται την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, αλλά δεν επιτρέπει απόλυτα την ελευθερία συνείδησης. Αλλά θα πρέπει να το διαβάσουμε στο σύνολο το Σύνταγμα. Η ελευθερία της σκέψης είναι εγγεγραμμένη πλέον στο Σύνταγμα. Και η βασική αρχή της έλλειψης των διακρίσεων, ανεξαρτήτως της αιτίας, είτε πίστης, είτε απόψεων κτλ, εγγράφεται πλέον στο Σύνταγμα και φυσικά και ο σημαντικότατο ρόλο του σεβασμού των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται πλέον στο Σύνταγμα. Και θα πρέπει ε, το Συνταγματικό Ανώτατο Δικαστήριο να ερμηνεύει τις διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν. Η κυριαρχία λοιπόν του διεθνούς δικαίου εγγράφεται επίσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εννοώ και, στο, και αυτό στο Σύνταγμα. Ο Υπουργό στην εισαγωγή αναφέρθηκε στα ειδικά χαρακτηριστικά τη ε, διαδικασία εκδημοκρατισμού του Μαρόκου. Πράγματι μέχρι την Αραβική Άνοιξη το Μαρόκο ήταν λίγο απομονωμένο. Αλλά η Αραβική αυτή Άνοιξη μας προσφέρει θα έλεγα νέου συμμάχου στην περιοχή και αυτό είναι το βασικό μάθημα. Σήμερα δηλαδή παράλληλα με τη διαδικασία τη μεταρρυθμιστική, την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το ρυθμό της, για τον αργό ίσως ρυθμό κτλ. Σήμερα όμως με τα κινήματα αυτά και ελπίζουμε και σε άλλες χώρες αδελφές να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα και να περάσουν σε πολιτικές αλλαγές ειρηνικές, έχουμε την δυνατότητα στη νότια πλευρά της Μεσογειακής Λεκάνης να προχωρήσουμε προς τη δημοκρατία. Ευχαριστώ κυρία Τζάμι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Μέχρι τις 4.30. Αν θέλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. οι παρεμβάσεις ε, των ε, φίλων με κάλυψαν σχεδόν ε, καθ' ολοκλήρου, δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Θα ήθελα μόνο να επιμείνω λίγο σε ορισμένα σημεία για να απαντήσω στις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τη Σαχάρα και τις συμφωνίες, فيها موضوع الصحراء εμείς δεν γνωρίζουμε καμία συμφωνία που να ε, διαπραγματεύεται αυτό το θέμα της Σαχάρας. Οι συμφωνίες που μας συνδέουν με την Ευρώπη αφορούν αμοιβαία συμφέροντα και ευρωπαϊκά και ε, μαροκινά και το ζήτημα, το πρόβλημα της Σαχάρας είναι πρόβλημα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και το Μαρόκο στενίζεται πλήρως ε, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζουμε δε οι ούροι άνεμοι του εκδημοκρατισμού που σήμερα πνέουν στις αραβικές ε, χώρες να έχουν θετική επίδραση και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης ελπίζουμε η πρόταση Αυτονομίας θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. يراعي مصالح المغرب ومصالح أوروبا ونأمل أن يعجل البرلمان الأوروبي بخروجه σε ό,τι αφορά τις γεωργικές συμφωνίες είναι θέματα αμοιβαίων συμφερόντων και αμοιβαίου ενδιαφέροντος ευρωπαϊκού και μαροκινού και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να επιταχύνει τις διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ελευθερίας του τύπου συγκεκριμένα, είναι γεγονός ότι πρόσφατα έγιναν κάποιες συζητήσεις σχετικά ε, και το νέο αυτό σύνταγμα σε ό,τι αφορά τις ελευθερίες και τα δικαιώματα ε, και τις λοιπές διατάξεις ε, του συντάγματος περί ελευθεροτυπίας, καθώς επίσης και το δικαίωμα στην πληροφόρηση, Όλα αυτά μας υποχρεώνουν όλους και τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να επανεξετάσουμε αυτά τα ζητήματα και να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που να εγγυάται με τρόπο αποτελεσματικό την ελευθεροτυπία. Euh, σε ό,τι αφορά λοιπόν το σχέδιο συντάγματος, θα αναζωογονήσει την πολιτική στη χώρα, θα τονώσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική και τη δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων. Οι κανόνες και οι διατάξεις του συντάγματος αυτού θα παροτρύνουν τους μαροκινούς πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και στις εκλογές προκειμένου. και οι Μαροκινοί πολίτες θα αποκτήσουν επίγνωση του γεγονότος ότι η ψήφος τους έχει βαρύτητα. Ε, θα μπορούν να επιλέγουν την κυβέρνησή τους ε, με βάση ένα πολιτικό και εκλογικό πρόγραμμα. Θα επιλέγουν για ποιον θα, θα ψηφίσουν και ε, αυτό θα επηρεάσει τη σύνθεση της κυβέρνησης. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες στο Μαρόκο γνωρίσαμε μια κατάσταση όπου παραμελήθηκε ο πολίτης και ε, απομακρύνθηκε από την πολιτική. Και ήταν χαμηλή η ε, συμμετοχή στις εκλογές. Ελπίζουμε επίσης, για να μην πω ότι είμαστε βέβαιοι, ότι το νέο αυτό σύνταγμα θα ενθαρρύνει και τους νέους να συμμετέχουν περισσότερο και να ψηφίζουν στις εκλογές. Η νέοι του Μαρόκου λοιπόν σήμερα θα πρέπει να περάσουν από την έκφραση της γνώμης τους μέσω των διαδηλώσεων σε μια ουσιαστική ε, συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι για το Μαρόκο η Ευρώπη ανέκαθεν ήταν στρατηγικός εταίρος στα σχέδιά μας και στα σχέδια εκδημοκρατισμού και στα σχέδια ανάπτυξης και παραμένει. Ένας εταίρος με τον οποίο ε, υλοποιούμε την πολιτική γειτονίας ο οποίος στη συνέχεια μας έχει παραχωρήσει αυτή την προηγμένη συνεργασία, αυτό το καθεστώς προηγμένης συνεργασίας και που τώρα πρόκειται να μας εχωρίσει το καθεστώς ε, ε του εταίρου στη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης ελπίζουμε να παραμείνουμε υπόδειγμα για τις χώρες της νότιας όχθης Μεσογείου προς ένα δημοκρατικό εκδημοκρατισμό με ειρηνικό τρόπο. Και σας υποσχόμαστε ότι δεν πρόκειται τώρα να επαναπαυθούμε σε αυτή τη συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλά ρητά θα εφαρμόσουμε το όσα λέει το Σύνταγμα, θα γίνει μια μεγάλη διαβούλευση για τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής και πάνω από 20 οργανικοί νόμοι θα ακολουθήσουν. Και άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή σας και την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ και τους φίλους οι οποίοι παρενέβησαν και έδωσαν απαντήσεις διαφορετικές μερικές φορές που εκπροσωπούν τις απόψεις που ακούγονται στη χώρα σας. Πράγματι ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας να αναγνωρίσουμε μια κατάσταση τόσο σύνθετη, αλλά νομίζω ότι οι στόχοι σας είναι οι ίδιοι με τους δικούς μας και θα μπορέσετε τους επόμενους μήνες με τη σωστή άσκηση της ηγετικής σας θέσης στον αραβικό κόσμο να οδηγηθείτε προς μια συνταγματική μοναρχία όπως θέλει να την καθορίσει ο, η αυτού μεγαλειώτης. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ε, ελπίζω σε λίγες μέρες να γιορτάσετε ένα βήμα προς τα εμπρός με το δημοψήφισμα το οποίο αποφασίσατε να οργανώσετε. Για μια ακόμη φορά καλώς ήλθατε και εις το επανειδήν.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 Ένα μικρό διάλειμμα πριν περάσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Πέντε λεπτά. Bene, allora cari colleghi, abbiamo atteso qualche minuto, ma abbiamo anche... Λοιπόν, θα μπορούσαμε να περιμένουμε λίγα λεπτά ακόμα, αλλά έχουμε αρκετά θέματα στη μερίσια διάταξη και πρέπει να ξεκινήσουμε έγκαιρα με την παρουσία του συνομιλητή μας, του κυρίου Νίκολας Westcott, ο οποίος είναι ε, διευθυντής ε, της E eh, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης υπεύθυνο για την Αφρική. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη συνάντηση τον Απρίλιο. Σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων θα συμμετέχει και ο κύριος Ντέβα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, ο οποίος θα φτάσει όπου να είναι και θα του δώσουμε το λόγο για να κάνει και αυτό στην εισαγωγή του σύντομα τώρα για να παρουσιάσω θα έλεγα το πώς έχουν τα πράγματα. Θα ακουστούν επίσης και κάποιες σκέψεις για την κατάσταση στην Δημοκρατία του Κόγκο. Έχουμε λίγες, λίγους μήνες για τις επόμενες προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο και δεν γνωρίζουμε αν θα οργανωθεί αποστολή παρατήρησης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κονγκό, στη Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα που έχουμε υπάρχουν κάποιες θα έλεγα εναλλακτικέ λύσεις και εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε με τα χρήματα τα οποία έχουμε το σύνολο των αναγκών. Υπάρχει επίσης το θέμα στο Σουδάν, το θέμα της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή του Αμπιέ και μετά οι τελευταίες εξελίξεις στο Νότιο Σουδάν, το οποίο προβλέπεται να ανακηρύξει την ανεξαρτησία του στις 9 Ιουλίου και σύντομα κατέληξε σε μια συμφωνία για τον ορισμό των συνόρων με το Σουδάν. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος Ντίβα θέλει να εισάγει ένα διαφορετικό θέμα πέραν αυτών στα οποία αναφέρθηκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντοτε είναι ευχάριστο να ε, μοιράζομαι την Προεδρία μαζί σας. Η χώρα αυτή χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από εμά όντως για να γίνει ένα έθνος από την αρχή και εγώ ήμουν ο εισηγητής στην έκθεση πριν δύο χρόνια για την δημιουργία ενός έθνους και ο ΙΕ ε, κατήρτισε μία επιτροπή το 2005 για την ε, ε, δημιουργία και τη δομή ενός έθνους και το Σουδάν αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλάβει κανείς τι είναι η ήπια εξουσία, soft power κατά τρόπον ώστε να μπορέσει ένα έθνος να αναλάβει ε, τη θέση του σαν ε, πλήρες ε, μέλος στην κοινωνία των εθνών και αυτό μεν ίσως δεν, δεν εφαρμόζεται πλήρως στο Νότιο Σουδάν αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε να επιδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να χορηγήσουμε την προστασία μας και να συζητήσουμε σαν ισότιμοι εταίροι με τον λαό του Νοτίου Σουδάν. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας και τώρα δίνουμε το λόγο ή στον εισηγητή μας. Κύριε Westcott, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά για μένα που επανήλθα. Θα είμαι σύντομος. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι οι ερωτήσεις σας. Θα ασχοληθώ λοιπόν με την κατάσταση ε, των φυλών στο Σουδάν ε, και θα θεωρήσω καταρχήν όπως είπε ο πρόεδρος ότι πλησιάζει η ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν στις 9 Ιουλίου κατόπιν του δημοψηφίσματος και όπου θα εκπροσωπηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τονίσουμε το συμβολισμό που αποδίδουμε σε αυτήν την εξέλιξη διότι συμμετείχαμε από την αρχή σε αυτή τη διεργασία. Η κατάσταση είναι πολύ πιο ευάλωτη από ό,τι ελπίζαμε όσο πλησιάζει αυτή η ανεξαρτησία. Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες υπάρχουν σοβαρές διενέξεις ή στο Αμπιέ και ή στο Κορταφάν και υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση αυτή ε, να χειροτερεύσει αντί να βελτιωθεί υπήρξε μία βαθμιαία επιδίνωση η οποία ξεκίνησε ε, με τον αποκλεισμό από τις βόρειες αρχές ε, των τροφίμων να φτάσουν στις διάφορες περιοχές του Νοτιού Σουδάν και υπήρξε ένοπλη ενεξή ε, και τέλος οι δυνάμεις του Σουδάν Σουδάν μπήκαν στο αμπιέ, εξεδίωξαν τους αντάρτες και τους πρόσφυγες. Έχουμε τώρα περί τις 100.000 προσφύγων που εγκατέλειψαν την περιοχή ε, του ΑΜΠΙΕ και άλλους πολλούς οι οποίοι έφυγαν από το νότιο Κορντοφάν προς, το, προς άλλες περιοχές και Τώρα ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία πολύ κακή κατάσταση ε, από πλευράς ε, ανθρωπιστικής στο Νότιο Κορδοφάν και γενικώ όλη την περιοχή. Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών ε, κρατών ο πρόεδρος Μπέκη επενεύει, ε, συμμετείχε στις διαβουλεύσεις και ο δικός μας εκπρόσωπος με δύο θετικές εκβάσεις. Καταρχήν εχθές υπεγράφει μία συμφωνία στην Αντίσα Μπέμπα μεταξύ της κυβερνήσεως του Νοτιού Σουδάν και της κυβερνήσεως ε, Βορείος του Καρτούμ για την τον αφοπλισμό του ΑΜΠΙΕ και για ε, μια ε, κατάπαυση του πυρός για να μπορέσει να διατηρηθεί η ειρήνη στο ΑΜΠΙΕ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να απομακρυνθούν από αυτό το σημείο. Ε, έχει υπογραφεί η συμφωνία αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί και ε, πρέπει οι ε, ε, διαμεσολαβητές να εξασφαλίσουν ότι σύντομα και οι αιθίωπες ότι σύντομα θα εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες και επίσης ο ε, μετά από παρέμβαση ε, του κυρίου Μπέκη στο νότιο ε, of υπήρξε μια κατάβευση του πυρός που αποφασίστη την Κυριακή και ο Αμπτελαζίδ Χιλού ο αρχηγός του SPLA στο νότιο Κορτοφάν συμφώνησε αλλά δεν υπάρχει κατάπαυση, μείωση προς το παρόν και ελπίζουμε ότι σήμερα θα υπάρξει μία προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και εκεί και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες αλλά ακόμη υπάρχει εκδίωξη πολλών προσφύγων, πολλοί εκδιώκονται από τα σπίτια τους και Γενικώ η κατάσταση προχωρά προς την διακήρυξη της ανεξαρτησίας 9 Ιουλίου και στη χρεσινή δήλωση η οποία ενδεχομένως ε, είναι κάτι που είδατε ε, συμφωνείται μία συλλογική προσέγγιση και ε, αναφέρονται όλες οι προκλήσεις και όλα τα μέτρα τα οποία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύουμε να αναλάβουμε για να ε, ενισχύσουμε την κατάσταση μεταξύ Βορρά και Νότου κατόπιν της ανεξαρτησίας και τι βοήθεια θα προσφέρουμε και στα δύο μέρη του Σουδάν στο μέλλον. Στο νέο Σουδάν θα συντονιστούμε με άλλους δωρητές, ιδίως τους ε, Νορβηγούς, τους Αμερικανούς, την ε, Παγκόσμια Τράπεζα και προσπαθούμε ε, να συνεννοηθούμε, να καταρτήσουμε τους τομείς όπου ο καθένας θα βοηθήσει διότι ξεκινάμε από το μηδέν και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ε, και να δούμε τι βοήθεια μπορεί ο καθένας να προσφέρει ε, θα υπάρξει μια αντιπροσωπεία μόλις υπάρξουν όλες οι αναγκαίες κυρώσεις και ε, θα υπάρξει ένας αρχηγός αντιπροσωπείας με βάση τη Τζούμπα. Ε, συμφωνήσαμε επίσης ε, για τη συνολική αντιμετώπιση της βοηθείας που θα προσφέρουμε στο Βόρειο Σουδάν για να υπάρξουν δύο βιώσιμα κράτη, διότι και τα δύο θα επιβιώσουν μόνο αν και τα δύο εξελίσσονται και αναπτύσσονται. Ε, στη βόρεια περιοχή την οποία ε, επισκεφθήκαμε τον προηγούμενο μήνα ξεκινήσαμε τις συζητήσεις και πάλι με τη κυβέρνηση του Χαρτούμ για να ε, επιληθούν τα διάφορα θέματα να μπορέσει να υπάρχει ξηρήνη στις παραμεθόριες περιοχές και να υπάρξει όμως πρόοδος και στον Ταρφούρ που παραμένει μία ανησυχία διότι η βία στον Ταρφούρ συνεχίστηκε φέτος και και τους τελευταίους 5-6 μήνες επιπλέον 70.000 άτομα έχουν ε, ε, μετατοπιστεί και ε, ενισχύουμε τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται στην Τόχα με τη, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Κατάρ και που οδήγησε στην υπογραφή μιας συμφωνίας πριν μία εβδομάδα στο τέλος Μαΐου και κατόπιν αυτού υπάρξει, υπάρχει μία βάση ε, για την κίνηση των ε, ανταρτών. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και ελπίζουμε ότι βασίζονται ε, το έγγραφο το οποίο έχει υπογραφεί. Και ερχόμαι στις μεγάλες λίμνες. Ευτυχώς η κατάσταση εκεί είναι λιγότερο εύθραυστη, ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά της χώρας, όπου εδώ πριν από λίγα χρόνια ε, ήταν ε, πολλές οι σειράξεις. Από ό,τι φαίνεται η ειρήνη κρατεί εκεί, γίνονται προσπάθειες φιλίωσης των διαφόρων ενόπλων ε, ομάδων που δρούν στην περιοχή. Μπορεί να μην προχωρούν γρήγορα, αλλά δεν οπισθοδρόμησαν κιόλας. Υπάρχουν κάποιες αργές κινήσεις σταθερές ε, η προσέγγιση Κιγκάλη-Κινσάσα φαίνεται να βαίνει καλώς και συνεργάζονται και οι δύο κυβερνήσεις. Η άμεση προτεραιότητά μας ε, σχετικά με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είναι να υποστηρίξουμε τις προετοιμασίες των εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου του 2011. 47 εκατομμύρια ευρώ υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα χρήματα αυτά ε, την Εφορευτική Επιτροπή, με την ε, Μινούσκο, την αντιπροσωπεία αποστολή του ΟΗΕ και άλλων, έτσι ώστε να ε, διεξαχθούν καλά οι εκλογές. Έχουμε αυτή την εβδομάδα μια διερευνητική αποστολή εκεί που θα μας αναφέρει μέχρι την άλλη εβδομάδα ως προς τις επιθυμίες και τις δυνατότητες, κατά πόσο θεωρείται σκόπιμο να αποσταλεί αντιπροσωπεία παρατήρηση εκλογών και η Ανεξάρτητη Εφορευτική Επιτροπή στην Κινσάσα αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσισεκέντη ε, θεωρούν ότι θα πρέπει να στείλει τέτοια αντιπροσωπεία παρατήρηση των εκλογών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ περιορισμένοι οι οικονομικοί πόροι και ε, έχουν πολλαπλασιαστεί οι εκλογές ε, που στέλνουμε αντιπροσωπεία παρατήρησης κυρίως στη Βόρεια Αφρική αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από κάποια κράτη-μέλη και είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι κάποιο είδου ε, παρατήρηση των εκλογών θα πρέπει να γίνει. Θα δούμε τώρα τι κλίμακα θα έχει αυτή, αλλά είναι απόλυτη ανάγκη να ε, αποσταλεί για να υποστηριχθεί ο λαός του Κονγκό στη μεταβασή προς μια ισχυρή και στεναρή δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη ε, αυτή η εκλογική αναμέτρηση γιατί είναι η δεύτερη και ε, αν πάνε καλά τα πράγματα θα δούμε ε, περίπου αντίστοιχη κατάσταση με την Ιγυρία που ο δεύτερος γύρος των εκλογών ήταν καλύτερος από τον πρώτο και ενισχύθηκε η δημοκρατία. αν πάει κάτι στραβά μπορεί να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση λοιπόν με πολύ ε, μεγάλο διακύβευμα. Μετέβησε η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό πριν από 15 μέρες είχα επαφές με στην αντιπολίτευση, η οποία ανησυχεί για τις προετοιμασίε για τις εκλογές. Μίλησα και με την Εφορευτική Επιτροπή και τον επικεφαλή, ο οποίο ήταν ε, ήσυχος και ικανοποιημένο από τη δουλειά που κάνουν. Ο εκλογικός νόμος ήταν αντικείμενο συζητήσεων όταν ήμουν εκεί και δέχτηκε διάφορα διαβήματα σχετικά. Στο μεταξύ έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και είναι πολύ καλύτερος από ό,τι θα περίμενε κανείς. Έγιναν ε, κάποιες αλλαγές. Ε, αποπειράθηκε η κυβέρνηση να αλλοιώσει το νόμο, αλλά αυτό απερίφθη στο Κοινοβούλιο. Είναι ενθαρρυντικό βήμα. Παρόλο που είναι πολύ σφιχτό το πρόγραμμα, η κατάσταση μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά ε, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι θα μπορέσει να διεξάγει τις εκλογές το Νοέμβριο η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και να προχωρήσει σε καλό δρόμο. Πάντως είναι ζωτική σημασία να συνεχίσουμε εμείς να συμμετέχουμε εκεί. Ε, γενικότερα συνεχίζουμε τα προγράμματα ε, οικονομικής ενίσχυσης και βοήθειας. Είχα την ευκαιρία να έχω μια επισκόπηση επιτόπου σύντομη παρόλο που η διακυβέρνηση παραμένει ζητούμενο. Έχουμε βρει πολλούς τρόπους πώς μπορούμε να δώσουμε αναπτυξιακή βοήθεια, να βοηθήσουμε δηλαδή το λαό της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό ε, για να κάνει τη διαφορά, ιδιαίτερα για το μέλλον και ιδιαίτερα για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια τάξη, με τη σεξουαλική βία και τη μεταρρύθμιση και των θεσμών. Βασικά είναι ζήτημα διακυβέρνηση όλα αυτά. Χρειάζεται ενίσχυση και της αποτελεσματικότητας των θεσμών αλλά και της διοικητικής μηχανής δηλαδή και της κυβέρνησης λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό για να είναι και περισσότερο υπόλογοι. Εκεί θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστώ κύριε Βέσκοτ. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ντανζό, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας. Τρία λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας σχετικά με το Σουδάν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα που άπτεται της πολιτικής και της ασφάλειας. Είναι μια διάσταση η οποία έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο στα πλαίσια του τρόπου που αντιμετωπίζεται το θέμα του Σουβάν. Και δεν εννοώ να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν ενδιάμεση ανάμεσα στο βορρά και στο νότο, αλλά προσπαθώντας να διασφαλίσουμε κάποιες ανάγκες του νοτίου Σουδάν, προσπαθώντας να λειτουργήσουμε σαν εκπαιδευτές. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι ευκταίο και πιστεύετε ε, εάν πράγματι οι εκπρόσωποι του Νοτιού Σουδάν θέλουν να εντάξουν αυτή την πλευρά της συνεργασίας μας. Για την δημοκρατία του Κονγκό, η αξιολόγηση την οποία κάνατε για τις δύο αποστολές που έχουμε επιτόπου, την αστυνομική και τη στρατιωτική, και ε, πράγματι ο ρόλος τον οποίο θα μπορούσε να παίξει η αστυνομική επιστολή στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας πιστεύετε ότι είναι κάτι το θετικό. Ευχαριστώ κύριε Ντανζό. Μπραντνερ τρία λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Westcoat. Έχω κάποιες ερωτήσεις αντίστοιχες με τις του κυρίου Ντανζό. πιθανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αστυνόμευση του αερολιμένα της Τζούμπα. Ποιος είναι ο στόχος της αποστολής, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Αστυνομία και πόσοι αστυνομικοί θα χρειαστούν και για πόσο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε το πρόγραμμά σας. Και δεύτερον, για το Κονγκό, θα μπορούσατε να είσαστε επακριβέστερος για την συνεργασία των δύο αυτών αποστολών. Πώς συνεργάζονται και σχετικά με το γραφείο της USR ε, που θα κλείσει στο τέλος Ιουνίου, οπότε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Είναι μια κατάσταση η οποία μας ανησυχεί και πώς θα αντιμετωπίσουμε την περιφερειακή διάσταση του γραφείου αυτού. Ευχαριστώ κύριε Μπράντερ. Κύριος Βότσον, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Σερ Βότσον επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι τρία λεπτά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Λυπάμαι που δεν ήμουν ε, εδώ στην αρχή της παρέμβασής σας, κύριε Westcott. Ε, η σχέση σας με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Είναι αλήθεια ότι θα κλείσουμε την υπηρεσία του και τι βήματα θα ληφθούν έτσι ώστε να διαβεβαιώσουμε τις, ε, τους πληθυσμούς της περιοχής ότι δεν θέλουμε απλά να απεμπλακούμε από εκεί. Ευχαριστώ κύριε Βότσον. Λόζινγκ τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εισαγωγή σχετικά με τις ε, εκλογές στο Κονγκό θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο για την διεξαγωγή διότι μιλήσατε για ε, μία αποστολή παρακολουθήσεως των εκλογών και θα ήθελα να ξέρω πώς η Επιτροπή σκοπεύει να στηρίξει την εκλογική διαδικασία οικονομικά ή υλικά και ε, ποιες είναι οι ε, διάφορες αποστολές που προβλέπονται ε, και επιπλέον εάν η, προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων ομάδων σχετικά με το Σουδάν, σχετικά με την δύναμη των 7.000 ατόμων, ξέρετε αν ορισμένα στρατεύματα έχουν ήδη ε, δεσμευτεί από τα κράτη για τις δυνάμεις του ΟΗΕ και αν ναι από ποια κράτη και ε, σχετικά με τη συμμετοχή πόσοι προβλέπονται. Ε, επίσης η δύναμη σε αυτή τι καθήκοντα θα αναλάβει. Προβλέπετε μία επέμβαση και στο Νότο που θα εδρεύει ή στα σύνορα ή σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή σε πολλαπλές περιοχές προβλέπετε εις το Νότιο Σουδάν μία ε, επέμβαση ή όχι ε, και εάν προβλέπεται συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα ήθελα να γνωρίζω τι ύψους και με ποιο στόχο. Σας ευχαριστώ εκ προημίου για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Βέσκοτ για την παρουσία του εδώ. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ εις ε, την RDC ε, και συμφωνώ σχετικά με ε, την εκλογική διαδικασία. Πιστεύω ότι έχει σωστά επιλεγεί η εκλογική διαδικασία σαν η κατάλληλη επέμβαση διότι πρέπει να υπάρξουν καλής ποιότητας εκλογές. Σχετικά με τον νότιο Σουδάν. Θα ήθελα να σχολιάσω και να υπενθυμίσω ότι όλοι χαιρόμαστε διότι τον ε, Ιανουάριο το δημοψήφισμα πήγε καλά αλλά είμαστε ε, κάπως ε, απογοητευμένοι διότι αυτή η διαδικασία είναι καθυστερεί και προβλέπεται ότι 9 Ιουλίου πρόκειται να υπάρξει η ανεξαρτητοποίηση. Οπότε ε, η ύπαρξη δύο βιωσίμων κρατών που θα ευημερούν είναι ένας ε, θαυμάσιο, ένα θαυμάσιο ψυχολόγιο, αλλά ρωτιέμαι αν θα υπάρχει κανένα ένα τέτοιο κράτος από τις 9 Ιουλίου και μετά. Διότι τι θα είναι το κράτος του Σουδάν μετά τις 9 Ιουλίου. Ε? Πέραν των ε, ενόπλων σειράξεων θα υπάρξει κράτος ουσιαστικό και δεύτερον, σχετικά με το Σουδάν, πώς εσείς ε, ε, αντιλαμβάνεστε την ε, επίσκεψη του Αλμπασίδη στην Κίνα που είναι μια χειρονομία σημαντική πολιτικά και θα ήθελα να έχω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη για τρία λεπτά. Είστε πάρα πολύ καλός, δεν θα το χρειαστώ. Μια ερώτηση έχω μόνο. Ε, στην υπόθεση του εμπορίου ε, ορυκτών ε, από τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό στις Πολιτείες προετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο για κρίσιμα νευραλγικά ε, μεταλλεύματα. Είναι το, ο νόμος Dodd Frank εσείς θα μπορούσατε να μας δώσετε τη γνώμη σας για την κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό και τι γίνεται με το εμπόριο σε αυτά τα μεταλλεύματα, ε, το προϊόν του οποίου χρηματοδοτεί οι αντάρτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να το κοιτάξει και να έρθει με αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βέστκοκ για την παρουσίασή του. Είχα την ευκαιρία να είμαι παρατηρητής εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στο Σουδάν αρχές Ιανουαρίου. Ε, είδα τις μεγάλες προσδοκίες και τον ενθουσιασμό του κόσμου για το δημοψήφισμα. Ταυτόχρονα όμως είχα και συνομιλίες με ε, τους ηθήνοντες στο Νότιο Σουδάν και εξέφρασαν φόβους και με τρόμαξαν και μένα ε, ότι ο δρόμος προς το μέλλον θα είναι δύσβατος. Όπως και οι γειτονικέ χώρες, ε, Σομαλία και ε, Τσάτ, και το Σουδάν θεωρείται ως αποτυχημένο κράτος και κινδυνεύει το νότιο Σουδάν να γίνει ένα νεοσύστατο αποτυχημένο κράτος. Όλοι εκεί οι άνθρωποι είναι ε, οι ενοπλοί πολέμαρχοι ε, από διάφορες φυλές που πολεμούν η μία την άλλη. Και δεν συμμετέχει ο απλός ε, πληθυσμός στα τεκτενόμενα και η μικρή υποδομή που υπάρχει διατηρείται στη ζωή από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να βοηθήσει ε, τη σύσταση του κράτους αυτού του Νοτίου Σουδάν και στο μέλλον και πώς έχει η συνεργασία με το Βόρειο Σουδάν γι' αυτό. Ε, και ουσιαστικά έχουν αγοράσει όλη την παραγωγή στο Νότιο Σουδάν οι Κινέζοι ε, και είναι και ο πρώτος εμπορικός εταίρος. Η Κίνα πώς συμπεριφέρεται στην περίπτωση αυτή και πώς αξιολογείται τη συμπεριφορά της. Έχουμε επαφές ως Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Τσέλερ. Η κυρία Ντεκεζέρ που τον προηγούμενο Ιανουάριο ήταν επικεφαλής της εκλογικής αντιπροσωπείας προς το Σουδάν και τον Νότιο Σουδάν. Παρακαλώ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι και πριν από δέκα μέρες και λιγότερο ήμουν στο Σουδάν. Βεβαίως χαιρετίζω τη συμφωνία που μόλις επετεύχθη για την περιοχή του ΟΑΜΠΙΑΙ. Ε, βέβαια, είναι και εύθραυστη όσο και περιορισμένη αυτή η συμφωνία. Αυτή ε, η συμφωνία θα ήταν κρίσιμη γιατί ε, πραγματικά τερματίζει τις μαζικές σφαγές του πληθυσμού, αλλά η διατήρηση της ειρήνης και ε, η διοίκηση είναι κοινή. Αλλά δεν ασχολείται συμφωνία καθόλου με την πολιτική διάσταση. Πού είναι τα σύνορα, πού θα νίκει, στο βορρά ή στο νότο. Πώς θα απεμπλακούν τα υπόλοιπα προβλήματα και θα απαγκιστρωθούν. Γι' αυτό έχω εγώ κάποια ερωτηματικά την παραμονή ε, ή τις παραμονές της ε, ανακήρυξης της ανεξαρτησίας. Αυτή η περιοχή του ΑΜΠΙΑ μέχρι τώρα ήταν ε, ένας κόμπος που εμπόδιζε διάφορα άλλα ζητήματα, ε, το πετρέλαιο, το νόμισμα, την ιδιότητα του πολίτη της χώρας, αλλά ήταν και ένα ατού που είχαμε εμεί στα χέρια μας και λέγαμε, εάν δεν συνεννοηθείτε, αν δεν τα βρείτε για αυτή την περιφέρεια, ε, ξεχάστε αυτά που μπορούμε να σας δώσουμε εμείς ως βοήθεια και για το Βορρά και για τον Νότο. Αυτή λοιπόν η διοικητική, στρατιωτική προκατακτική συμφωνία. Από εμά, πώς αξιολογείτε, πώς θεωρείτε ως ε, χειρονομία καλής θέλησης εκατέρωθεν και θα μπορέσουμε να συνοδεύσουμε αυτά τα δύο κράτη ή μήπω θα τους ζητήσουμε και περισσότερα. Δηλαδή επιτέλους να αποφασίσουν και για τα υπόλοιπα σημαντικά προβλήματα που παραμένουν εκκρεμοί. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Διότι Εάν ε, αφήσουμε αυτό το χαρτί τώρα από τα χέρια μας δεν θα έχουμε άλλο μέσο πίεσης. Και είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο που συνδέεται, επίκειται και δημοψήφισμα κανονικά στην περιοχή του Αμπέη και ε, σε άλλες περιοχές εκεί. Τι θα γίνει αυτό, θα παγώσει, θα το εγκαταλείψουμε, θα το πεμπολίσουμε, θα το χάσουμε. Και μια ερώτηση προς τους συναδέλφους που προβληματίζονται μήπως είναι αποτυχημένη χώρα από την αρχή της, ε, το Νότιο Σιδά. Εδώ και ένα χρόνο και πλέον από τις εκλογές του 2010 και μετά ζω μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Σουδάν και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι τους είδα να κάνουν θαύματα και οργανωτικά και τεχνικά και πολιτικά. Τη στιγμή που θεωρούσαμε ότι όλα πάνε χαμένα, κάτι γίνεται και ξαναπαίρνει μπρο. Υπάρχει ε, μια τρομερή θέληση, ένας διακαής πόθος στο Νότιο Σουδάν να αποκτήσουν κράτος. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει κανένα θεσμό, ούτε σχολείο, ούτε δρόμο, ούτε νοσοκομείο, ούτε τίποτα και μεγάλη κίνδυνη για διαφθορά. Αλλά, έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε Μακρύγορο, δεν θα ήθελα από τώρα να κινδυνολογήσω κι εγώ Κασάνδρα ότι θα αποτύχει από χέρι χώρα ε, και να απεμπολίσουμε αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ κύριε Ντεκάιζερ. Κλείνει τη συζήτηση ο συμπρόεδρος μας ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πριν περάσω στα συμπεράσματα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Βότσον για το ότι πήρε το παράσημο της, ε, αυτού μεγαλειότητας της Βασιλίσης και είναι πλέον Σερ Βότσον. να ρωτήσω, να θέσω κάποιες ερωτήσεις στον Νίκλα Σόκλε για το Κονγκό. Πριν λίγους μήνες είχαμε μία συνάντηση στα πλαίσια των ΑΚΕ στο Κονγκό και περάσαμε το ποτάμι και πήγαμε και στον Κονγκό Μπραζαβίλ. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Σασού και ανησυχούσε ο πρόεδρος ε, του Κονγκό Μπραζαβίλ για το κύμα των προσφύγων από τη Δημοκρατία του Κονγκό που ερχόντουσαν στη Δημοκρατία του Κονγκό Μπραζαβίλ. Αν οι εκλογές δεν πάνε όπως εμείς περιμένουμε ότι θα πάμε, αυτό θα του δημιουργήσει προβλήματα, φοβάται ο πρόεδρος του Κονγκό Μπραζαβίλ. Δεν ξέρω αγαπητέ Νίκολας αν έχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται και ελέγχεται μάλλον η κατάσταση Και τι γίνεται με τους πρόσφυγες, οι πρόσφυγες θα ψηφίσουν, θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Θα κάνουμε ό,τι είχαμε κάνει στο Μπαγκλαντές παλιότερα και στο Πακιστάν όπου ελέγχεται η συμμετοχή τους σε πάση περιπτώσει. Η δεύτερη ερώτηση Κάτι το οποίο παρατήρησα όταν πήγα και στις δύο χώρες με τον Μακονγκό, ότι δεν έχουν δρόμους ουσιαστικά. Έχουν όμως ένα πυκνότατο σύστημα ποταμών για τις μεταφορές. Δεν έχουμε βοηθήσει καθόλου τις μεταφορές ε, σας, τις παραποτάμιες. Είναι πολύ εύκολο να τους βοηθήσουμε νομίζω. Δεν ξέρω αν κάποιος από την γραμματεία σας ή από την υπηρεσία σας εξετάζει το θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς θέλετε να απαντήσετε σε αυτά, θέλετε να περάσω στο να κλείσω τη συζήτηση ή τι ακριβώς θέλετε. Θα πρέπει να απαντήσετε πρώτα μάλλον. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να επανέλθω στις ερωτήσεις που τέθηκαν και θα ξεκινήσω με το Σουδάν. Τέθηκαν ερωτήσεις λοιπόν για την ε, στήριξή μας στον τομέα της ασφαλείας στο Νότιο Σουδάν. Στα πλαίσια της κατανομής των ευθυνών για τη βοήθεια προς τον Νότιο Σουδάν, ο τομέας της ασφαλείας είναι ένας τομέας στον οποίο θα ηγείται η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά φυσικά θα ήθελε να βοηθηθεί από άλλες δωρήτριες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη σε ορισμένου τομεί, την οποία θα θέλαμε να είμαστε προθυμότατοι να θέσουμε στη διάθεση της κυβέρνησης του Νοτιού Σουδάν όταν αυτό κριθεί κατάλληλο. Συζητήσαμε επίσης και μια ολόκληρη γκάμα δράσεων σε τρεις βασικούς τομείς. Η συζήτηση στο Συμβούλιο χτες ε, δείχνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά. Ο πρώτος τομέας είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του αεροδρομίου της Τζούμπα. Το αεροδρόμιο της Τζούμπα για όσους πήγαν είναι ένας πάρα πολύ απλός χώρος και θα δυσκολευτεί να υποδεχθεί όλους τους αρχηγούς κρατών την 9η Ιουλίου και φυσικά θα πρέπει να είναι υπεύθυνο από τις 9 Ιουλίου και για τον εναέριο έλεγχο. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις λοιπόν και μιας και είναι μια χώρα η οποία ξέρετε ότι δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα θα εξαρτηθεί ιδιαίτερα από τη χρήση του αεροδρομίου της. Η ασφάλεια λοιπόν του αεροδρομίου είναι πάρα πολύ σημαντική εφόσον θέλουμε να υπάρξουν τακτικές ε, εμπορικές πτήσεις γιατί αλλιώ οι εταιρείε δεν θα πάνε σε, ε, μια, σε, ένα αεροδρόμιο στο οποίο δεν υπάρχει ασφάλεια. Εδώ έχουμε εμπειρογνωμοσύνη και μέσω του Eurocontrol γνωρίζει πως λειτουργούν τα πράγματα και θα μπορούσαμε να το προσφέρουμε αυτό σαν ε, τεχνική βοήθεια. Επίσης, ένας άλλος τομέας, στον οποίο έχουμε μια κάποια εμπειρογνωμοσύνη, είναι οι παραποτάμιες συγκοινωνίες και εφόσον επίσης υπάρχει η δυνατότητα να βοηθήσουμε και στο θέμα της ασφάλειας των σύνορων. Για πάρα πολύ καιρό, στα σύνορα βορρά-νότου, στην ουσία η λογική οδηγεί ε, σε αυτό το οποίο θα ονομάζαμε ένα soft border, δηλαδή ε, όχι αυστηρά ελεγχόμενες ε, όχι αυστηρά ελεγχόμενα σημεία διαβα, δια, δια, περάσματος από το ένα μέρος στο άλλο, ιδιαίτερα με ένα ομαδικό πληθυσμό, ένα τέτοιο σύστημα soft border θα μπορούσε πράγματι ε, ένα σύστημα ήπιων τελωνιακών ελέγχων, εν πάση θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Όλα αυτά βέβαια είναι αντικείμενο συζήτηση με τα κράτη-μέλη, ακούγονται συζητήσει, ακούγονται προτάσεις, δεν έχουμε όμως συγκεκριμένα προγράμματα, δεν έχουμε συζητήσει όλα τα προγράμματα αυτά. Υπάρχουν πάντως δυνατότητες ε, με τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε τον Νότο. Ο κύριος Πρέντα είπε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ε, στην δημιουργία δύο πραγματικά χωρών βιώσιμων ε, βιώσιμων και ε, με τη δυνατότητα να ευημερήσουν. Μέχρι τώρα είχαμε ένα κράτος το οποίο δεν ήταν βιώσιμο γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να έχει την εσωτερική συνοχή και οι πληθυσμοί της χώρας αποφάσισαν να δοκιμάσουν ε, τις δύο χώρες. Δεν έχουμε εγγυήσει για το ότι θα πετύχει κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι και τα δύο αυτά κράτη θα πετύχουν εφόσον και τα δύο ε, είναι θα έλεγα βιώσιμα. Φοβάμαι ότι αν αποτύχει ένα από τα κράτη αυτά θα αποτύχουν και τα δύο. Θα αποτύχει και το άλλο. Απαιτείται λοιπόν να βοηθήσουμε με σωστό τρόπο και τον Βορρά και τον Νότο. Προσπαθούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ε, τις χώρες αυτές Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το Σουδάν και για το Νότιο Σουδάν ότι έχει αποτύχει, οπότε δεν είναι ακόμα κράτος κανονικά, οπότε πώς να αποτύχει εφόσον δεν είναι κάτι. Αλλά πάντως αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παραδεχτούμε ότι η οργάνωση SPNN στην ουσία έχει λειτουργήσει συνεκτικά για την χώρα η κυβέρνηση δεν είναι αποκλειστική βέβαια του σχηματισμού αυτού και το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό έτσι ώστε να είναι αναπόσπαστο τμήμα του κράτους, το SPNN και όχι ε, θα έλεγα το ίδιο το κράτος. Η διαδικασία θα είναι μακρά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού του Νότου που πηγαίνει στο SDLA και οι δωρητές στην ουσία υποστηρίζουν οικονομικά ε, την υγεία, την παιδεία κτλ. Θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα βέβαια και όσο νωρίτερα μπορούμε να περάσουμε στις αλλαγές αυτές, τόσο νωρίτερα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες δομές και δομές οι οποίες να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του λαού τέθηκε επίσης ένα θέμα σχετικά με το αμπιέ. Η συμφωνία που υπεγράφει χθε από το αμπιέ στην ουσία αποκαθιστά το status quo που ισχύει πριν από την πρόσφατη κατοχή από δυνάμεις του Βορείου Σουδάν δεν μας φέρνει πιο γρήγορα στην επίλυση του προβλήματος και των μεθοριακών προβλημάτων τα οποία υπάρχουν. Κατά κάποιο τρόπο την καθιστά ακόμα πιο δύσκολη. Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε και σε ένα δημοψήφισμα. Αλλά εφόσον έχουν εκδιωχθεί οι κάτοικοι του Σαμπιέ, είναι δύσκολο να κάνουμε δημοψήφισμα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την κατάσταση. Οι δυνάμεις που υπάρχουν εκεί αντιπροσωπεύονται σε τρία επίπεδα θα έλεγα. Υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας στο Σουδάν, υπάρχει η UNOMED η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο και καθορίζεται, θα πρέπει η εντολή να ανανεωθεί μάλλον σύντομα και θα δούμε τι θα γίνει ε, μετά την ανεξαρτησία του Νότου. Δεύτερον, σύμφωνα με τη συμφωνία θα υπάρξει μια νέα δύναμη εφιοπικού στρατού με την καθοδήγηση και την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών που θα τηρήσει την τάξη στο ΑΜΠΙΕ. Και οι Βόρειοι και οι Νότιοι έχουν συμφωνήσει να επιτρέψουν τους Αιθίωπες μόνους να προχωρήσουν στην επιβολή της τάξης. Υπάρχει δηλαδή η αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών θα υπάρξει μια εντολή των Ηνωμένων Εθνών για να προχωρήσουν οι Αιθίωπες. Και τρίτον, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα ε, βοηθήσουν ε, την κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάμ να αποκαταστήσει, ε, να μετατράψει το SPLA σαν παράδειγμα σε τακτικό στρατό κτλ. Τώρα ο ρόλος της Κίνας στο Σουδάν. Η Κίνα θα είναι παρούσα, δεν έχουν βέβαια πάρα πολλές επενδύσεις στο Νότιο Σουδάν όπως έχουν στο Βορρά, ενδιαφέρονται όμως και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε μαζί τους γιατί η σταθερότητα της περιοχής είναι πολύ σημαντική και για αυτούς όπως είναι και για εμάς ανακοίνωσαν ότι θα καλέσουν τον πρόεδρο Μπασίρ να επισκεφθεί την Κίνα. Η Ένωση θεωρεί ότι μια χώρα την οποία επισκέπτεται ο πρόεδρος Μπασίρ εφόσον είναι μέλος ε, της συνθήκης της Ρώμης θα πρέπει να συλληφθεί και να υπάρξει παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση θα έλεγα. Τώρα για τη δημοκρατία του Κονγκό. Εκεί έχουμε δύο αποστολές, η μία αστυνομική, η μία στρατιωτική και οι δύο συνεχίζουν τις εργασίες τους και οι δύο είναι επιτυχείς, θεωρούνται επιτυχείς. Προσπαθούμε να δούμε τις συνέργειες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο αυτές αποστολές συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους των ομάδων αυτών. Δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει στην πρόταση να συμπτύξουμε τις δύο αυτές ομάδες. Θα δούμε. δεν, οι επιτυχίες δεν ήταν στιγμιαίες των προσπάθειών μας εκεί και γι' αυτό θα πρέπει σταδιακά να συνεχίσουμε να τις αξιολογούμε για να δούμε αν θα συνεχιστεί η λειτουργία του στο μέλλον. Τώρα για το ρόλο του ειδικού εκπροσώπου στην περιοχή των λιμνών. Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό γιατί ίσως να υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Είχαμε με τον τελευταίο εκπρόσωπο έναν μια εξαιρετική προσωπικότητα που ήταν στη θέση μέχρι τον Ιανουάριο. Πήγε τόσο καλά που έγινε αρχηγός της αντιπροσωπείας μας στην Νότια Αφρική. Από τότε, από τον Ιανουάριο, υπάρχει μια προσωρινή απουσία ειδικού εκπροσώπου για την περιοχή των λιμνών. Αυτό συνέπεσε και με τη δική μου έλευση και γι' αυτό πρότεινα να επανεξετάσουμε τις επιλογές που έχουμε να ορίσουμε ένα νέο εκπρόσωπο, να σταματήσουμε να έχουμε ειδικό νέο εκπρόσωπο, ειδικό εκπρόσωπο και να αντιμετωπίσει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, τις αποστολές τις οποίες αναλάμβανε ο ειδικό εκπρόσωπος. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η κατάσταση εν μεταξύ έχει αλλάξει και στο Κονγκό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Δημοκρατία του Κονγκό, Κινσάσα, η κατάσταση είναι πιο σταθερή από ό,τι ήταν τότε όταν διορίστηκε ο ειδικό εκπρόσωπος εδώ και 10 χρόνια. Τότε υπήρχε ένας ενεξελίξη εμφύλιος. Αυτό δείχνει και την πολύ καλή δουλειά βέβαια που έκανε ο ειδικό εκπρόσωπος και όλων των εμπλεκομένων Υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, υπάρχει αυτή τη στιγμή επικοινωνία ανάμεσα στην Κινσάσα και την πρωτεύουσα της Ρουάντα και η κατάσταση είναι πιο σταθερή, αν και εύθραυστη βέβαια σε σχέση με το παρελθόν. Δεύτερον, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, την οποία δεν είχαμε στο παρελθόν. Όταν χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι σε ένα διεθνές πρόβλημα έπρεπε να ορίσει ένα ειδικό διαμεσολαβητή εκπρόσωπο. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Έχουμε την ύπατο εκπρόσωπο για την εξωτερική δράση και έχουμε πλέον τα μέσα να λειτουργήσουμε και σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν προσπάθειες που γινόντουσαν από τον ειδικό εκπρόσωπο που ήταν διαμεθοριακές, αντιπροσώπευαν την περιφερειακή μας παρουσία θα έλεγα εκεί και όχι στο εσωτερικό μία συγκεκριμένη χώρα. Και γι' αυτό συζητάμε ορισμένες προτάσεις για να μπορέσουμε να συμπτύξουμε τις αποστολές του ειδικού εκπροσώπου με την δράση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και της αντιπροσωπείας που έχουμε εκεί. Αυτό θα απαιτήσει κάποιους ειδικού πόρους που θα μεταφερθούν από το γραφείο του ειδικού εκπροσώπου στο γραφείο της αντιπροσωπείας μας εκεί. Και αντί να έχουμε λοιπόν ένα νέο ειδικό εκπρόσωπο, θα ορίσουμε ένα συντονιστή από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο οποίος θα διασφαλίσει να υπάρξει συγκέντρωση ακριβώς της περιφερειακής διάστασης της προσπάθειας και να υπάρξει μια ενιαία ομάδα η οποία να ασχολείται με τα θέματα αυτά και να συντονίζει τις δραστηριότητες των αντιπροσωπιών στην περιοχή και όχι δύο ομάδες, μία της εξωτερικής δράσης και μία του ειδικού εκπροσώπου. Θέλουμε να τα εντάξουμε όλα αυτά λοιπόν στο εσωτερικό της εξωτερικής δράσης. Έχουμε δυσκολίες, αντιμετωπίζουμε ένοπλες συμμορίες, παράνομο εμπόριο ορυκτών, βία, βία σεξουαλικής μορφής επίσης και δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν οι προσπάθειές μας. Αυτές είναι οι προτάσεις πάντως που θα γίνουν χοντρικά σύντομα. Για το θέμα των ορυκτών, που, των παρανόμως διακινουμένων. Το εξετάζουμε το θέμα, συνειδητοποιούμε το φαινόμενο, έχουμε και τη διαδικασία του Κιγκάλη, η οποία δόξα τω Θεώ δουλεύει καλά Βέβαια την επιτυχία την οποία, στην οποία έχουμε φτάσει μέχρι τώρα σε ένα συγκεκριμένο ρηκτό δεν μπορούμε να την επαναλάβουμε σε όλα. Για να μπορέσουμε αποτελεσματικοί απαιτείται να έχουμε στη διάθεσή μας έναν μηχανισμό ο οποίος τελικά θα αποβεί αντιπαραγωγικός. Εξακολουθούμε να εξετάζουμε το θέμα, να δούμε τι θέλουν οι Αμερικανοί να κάνουν σε νομοθετικό επίπεδο αλλά οι συζητήσεις που έγιναν μέχρι τώρα είναι ότι μιας και είναι τόσα διαπερατά τα σύνορα όπως σήμερα και αν δεν έχουμε μια συγκεκριμένα ελεγχόμενη αυστηρά αγορά είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιο φάρμακο ε, και πράγματι ένας τέτοιο μηχανισμός θα είναι ιδιαίτερα ακριβώς και θα στο τέλος θα αποβεί μη χρήσιμος. Έχουμε βρει λοιπόν κάποιους τρόπους θέλουμε να εμποδίσουμε το παράνομο εμπόριο των ρηκτών αυτών που οδηγούν στη χρηματοδότηση παρανόμων ενόπλων ομάδων. Θέλουμε να αποκατασταθεί πλήρης τάξη δικαίου στην δημοκρατία του Κόγκο. Αυτή είναι φυσικά η βασική, η βασική προοπτική μας. Αν το πετύχουμε αυτό σχετικά γρήγορα και αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό. Και τέλος για την εκλογική διαδικασία. Υποστηρίζουμε με 2 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν απατώ, με την ασφάλεια των εκλογών για τη διεξαγωγή τους αυτή καθ' αυτή. Για να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ειρηνικό και συνεργάσιμο θα πρέπει να αποφύγουμε μεταναστευτικά ρεύματα και ρεύματα προσφύγων. Γι' αυτό ανησυχεί ο πρόεδρος Ασούγκεσο της Δημοκρατίας του Κονγκό Μπραζαβίλ. Ε, προς το παρόν ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και επαναλαμβάνω είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ε, δεινά. Σε ό,τι αφορά τις ποτάμιες μεταφορές βεβαίως είναι λογικός αυτός ο δρόμος και θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε θα το συστήσω με τους συναδέλφους μου που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης. Αφήστε δε που έχει ήδη προβλεφθεί. Και υποστηρίζουμε ένα έργο, εξετάζουμε 40 εκατομμύρια ευρώ περίπου, αλλά δεν έχουν όλα αυτά ακόμα ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνοκ ζήτησε το λόγο, αφού ε, είχα ήδη δώσει το λόγο στον κύριο Γουέστον. Ένα λεπτό, ένα λεπτό πρόεδρε. Ε, γεια σας κύριε Γουέστον, χαίρομαι που σας βλέπω. Ενδιαφέρον αυτό το θέμα για τα διαμάντια του αίματος που είδαμε στον τύπο ότι διαμάντια από Τη Ζιμπάμπουε ανακατεύονται ε, με νόμιμα διαμάντια και μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ξέρετε εσείς. Και εσείς πιστεύετε ότι η Λιβύη, ε, μάλλον ότι το Σουδάν μπορεί να είναι λύση για τον Κατάφη και να πάει να βρει εκεί ε, στη Χαρτούμ το φίλο του τον Μπασίρ που είναι και αυτός υπόδικος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης μου είπαν ε, ε, ιδιαιτέρως ότι πρόκειται να αναγνωρίσουν το Σομάλιλαντ ως ανεξάρτητο κράτος. Και τι θα γίνει αυτό και άλλες χώρες της Αφρικανικής Ένωσης θα συνεχίσουν και αν το πράξουν αρκετές χώρες μήπως ε, μπουν στον πειρασμό και ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ λοιπόν. Έχετε κύριε Βέσκοπ το λόγο να απαντήσετε πολύ σύντομα και στα τρία θέματα. Συζήτησα για την διαδικασία του Κίμπελι όταν ήμουνα προσφάτως στην Νότιο Αφρική και υπάρχουν ψήφεροι ότι υπάρχει μία συζήτηση για τη διαδικασία του Κίμπελι στην Κινσάσα. Συζητούνται τα θέματα αυτά, δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Δεύτερον, δεν είναι κάτι στο οποίο εγώ μπορώ να υπολογίσω πού θα καταλήξει ο κύριος Καντάφη. Αφήνω αυτό το θέμα σε άλλους. Αλλά όσον αφορά την ε, αναγνώριση του Σομάλιλαντ ε, άκουσα ότι το Νότιο Σουδάν ε, σκοπεύει να το αναγνωρίσει και πιστεύω ότι δεν είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβερνήσεως η οποία έχει πολλά πιο σημαντικά θέματα και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διάφορα προγράμματα προγράμματα στην περιοχή Σομάλι Λαντ και ο, ο πρόεδρος ενδιαφέρεται ε, αλλά η θέση μας όσον αφορά την ακαιρεότητα του κράτους της Σομαλίας δεν είναι κάτι το οποίο θα αναθεωρήσουμε. Αν ή αλλάξει άποψη θα το ξανασυζητήσουμε αλλά θα δούμε αν η Αφρικανική Ένωση με συγχωρείτε αλλάξει άποψη. Ευχαριστώ. Ε, τώρα εγώ έκανα την αρχή και ο συμπρόεδρος κύριος Ντέβα θα καταλήξει. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι ε, και θα είμαι σύντομος. Πιστεύω ότι ακούσαμε ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα για μια σημαντική περιοχή, για, για δύο σημαντικές περιοχές οι οποίες είναι σημαντικές για μας και έχουν πρώτες ύλε που είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάπτυξη. Η συνεργασία που έχουμε και με την DRC και με το Κονγκό Μπραζαβίλ και με το Βόρειο και Νότιο Σουδάν είναι σημαντικές ε, και υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτών των χωρών που είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό και πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε διακηρύξει το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, η Επιτροπή μας προσπαθεί να προωθήσει τη δημιουργία εθνών και τη δημιουργία καλών ε, εταιρικών σχέσεων που θα ε, καταλήξουν σε ανάπτυξη για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτά. Ακούσαμε λοιπόν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα και τελειών, φεύγοντας από αυτή τη συνεδρίαση δεν ξέρω πόσο θα έχουμε τον πρόεδρο Μπασίρ από τη μία πλευρά και πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί με την κυρία Άστον από την άλλη όταν και οι δύο θα αναλάβουν τα κυρίαρχα καθήκοντά τους στις 9 Ιουλίου ε, και εάν δεν καταφέρουν ε, να τους ε, έχουμε ε, χωριστά εκτός από ενδεχομένως μία κοινή φωτογραφία. Δεν θέλουμε η κυρία Άστο να καταλήξει στο δικαστήριο της Χάγης μαζί με τον συμφωτογραφόμενό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν. La nostra Διάλειμμα λοιπόν και μετά θα συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες.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 Σας καλώ να βάλετε τις ε, κάρτες σας εις ε, το μηχάνημα και να ελέγξετε αν τις έχετε μαζί σας. Και πριν ξεκινήσουν οι εργασίες σας θέλω να συγχαρούμε τη συνάδελφο Άουταλα Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία στην οποία θα πάρει μέρος στις εργασίες της Επιτροπής μας γιατί έγινε υπουργό. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την συνεργασία της μαζί μας. Ιδιαίτερα παραγωγική, ιδιαίτερα ευαίσθητη παρουσία της και ε, πράγματι και όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εν πάση περιπτώσει. Ε, και την ευχαριστώ για την προσπάθεια την οποία κάναμε από κοινού. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Τώρα στο πρώτο θέμα αφορά την έκθεση τη σχετική, ε, μάλλον την έκθεση Τόκες. πολιτική προστασία, ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πριν από την ψηφοφορία έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Μπρέντερ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να ζητήσω στην τροπολογία 7 τη δική μας ψηφοφορία κατά τμήματα. Γιατί το πρώτο τμήμα αναφέρεται στο μέσο σταθερότητας και το δεύτερο αφορά κάποιες αποστολές Πά, αλλά να είναι ξεχωριστές. Ε, δεν μπορούσαμε να το καταθέσουμε ξεχωριστά γιατί είναι η ίδια παράγραφος. Ε, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ότι η αντιμετώπιση των κρίσεων και των θεομηνιών δεν είναι στη νομική βάση του μέσου σταθερότητας και δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ στην τροπολογία. Θα βοηθήσει λοιπόν η ψηφοφορία κατά τμήματα για να διορθώσουμε την κατάσταση και να μπορέσουν οι βουλευτές να ε, ψηφίσουν για το δεύτερο τμήμα. Ευχαριστώ. Μου είπαν ότι συμφωνεί ο εισηγητής, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από πλευράς μου και γι' αυτό θα προχωρήσουμε τώρα. Ε, με ξεχωριστή ψηφοφορία στο 7. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 3 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 4 υπέρ, Θέλετε ηλεκτρονικός έλεγχος να γίνει για την 3. Καλώς. Ξεκινάει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 3. Πέρα στις ψηφοφορίες. 30-21 και εγώ. Ε, ψήφισα κατά και η κυρία Γιαννάκου, οπότε απερίπτεται. Λοιπόν, τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Έχει αποσυρθεί η έκτη. Έχουμε σε τρία τμήματα την ψηφοφορία της 7. Σε δύο τμήματα μάλλον την 7. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Η 8. Ναι, η 8 λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 9 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Η 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο, μου φαίνεται ότι απερίφθη, αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 14 ξεκινάμε. Και θα συμπληρώσουμε τις ψήφους. Α, ε, εντάξει, έχει την κάρτα της κυρία Γιαννάκου. Λοιπόν, πέρα στις ψηφοφορίες. 33 λοιπόν, κατά 23 υπέρ, 15 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 17 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική ψήφος τώρα για το σύνολο της γνωμοδότησης. Ξεκινάμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 53 υπέρ με 2 κατά και μηδέν αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή τον κύριο Τόκες. Περνάμε τώρα στον κανονισμό που εφαρμόζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Η 14 απεσύρθη με την 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 16 Α, θέλετε ηλεκτρονικός έλεγχος να υπάρξει για τη 15. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 25 υπέρ κατά Αποχές. Απερίφθη. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 29 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή έχει γίνει δεκτή 31 λοιπόν περνάμε τώρα στην 32 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 33 υπέρ κατά Αποχές. Απερίπτωται. 34. Προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 7 γίνεται δεκτή. Η 35 όχι. Η 8 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 37 υπέρ. Αν θέλετε να υπάρξει για την 36 ηλεκτρονικό έλεγχος λοιπόν. Είδα το βλέμμα σας, δεν φανήκατε σίγουροι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμο αυτό που κάνουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, α εγώ ψηφίζω κατά, 27-27 λοιπόν, Α, συγγνώμη, πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση. Μου λέγουν ότι η ψήφος ε, του Προέδρου ισχύει και απορρίπτεται. Αλλά καλά κάνατε που ζητήσατε παλήθες. 37 λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 9 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 10 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 38 και η 39 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 38 και 39 λοιπόν. Πέρα στις ψηφοφορίες. 25 κατά, 31, 32 υπέρ μάλλον, 24 κατά, δεκτή. Περνάμε στη 12 τώρα. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 12 παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Λοιπόν, αυτό ήταν ξεκάθαρο. 47 υπέρ, 7 κατά. Λοιπόν, με μεγάλη πλειοψηφία. 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονική ψήφος για το σύνολο τώρα. Ψηφίζουμε. Κάποιοι δεν έχουν ψηφίσει. Έβαλαν την κάρτα τους αλλά δεν ψήφισαν κάποιοι. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία από την αρχή. Τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίζεται εκ νέου για το σύνολο, γιατί υπήρξε ένα πρακτικό πρόβλημα τεχνικό. Μόνο δύο δεν ψήφισαν με την κάρτα τους λοιπόν, πέρα στις ψηφοφορίες. 49 υπέρ, ένας κατά και 5 αποχές. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν υπέρ ε, του εισηγητή συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε πριν την επόμενη ψηφοφορία θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ κατηγορηματικά κατά της διαδικασίας που νομίζω και είναι και παράτυπη ε, για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΕΠΑ. Γι' αυτό θα καταψηφίσουμε όλες τις παραγράφους. Διαμαρτύρομαι εντονότατα. Μπορώ να σας παραθέσω και ολόκληρο κατάλογο αντιδημοκρατικών ε, διαδικασιών και συμπεριφορών, αλλά το αφήνω στην άκρη. Νομίζω τα γνωρίζετε και μόνο σας διαμαρτύρομαι και αντιτίθεμαι στη διαδικασία αυτή και παρακαλώ να εγγραφούν όλα αυτά στα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Καζίνη. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι έχω κάποιες απορίες. Έχουμε να κάνουμε με ένα ψήφισμα το οποίο αφορά τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις και η ΑΦΚΟ, η Επιτροπή μου, έχει αρμοδιότητες επ' αυτού. Οπότε θα έπρεπε από κοινού να το συζητήσουμε το θέμα. Εδώ μου λένε ότι το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το θέσω στην Πολωνική Προεδρία, γιατί αυτή ασχολείται με το θέμα των σχέσεων με τα κοινοβούλια. Εν πάση περιπτώσει εκφράζω κάποιες ανησυχίες και εγώ λοιπόν εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής μου Επιτροπής. Ευχαριστώ, ο κύριος Μπροκ. Και είδα και τον κύριο Βανόρντεν μετά. Θα ήθελα ε, καταρχάς να συμφωνήσω με τον κύριο Κασίνη ότι οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις θα πρέπει να συζητώνται και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αλλά εμείς μιλάμε τώρα εδώ για την ΚΕΠΑ και για την ΕΠΑ. Αυτό είναι αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Δεν έρχεται σε καμία αντίφαση και είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε. Και το θέμα αυτό μέχρι τώρα σε τούτη εδώ την Επιτροπή το διαπραγματευόμαστε. Ευχαριστώ. Κύριε Βαν Ευχαριστώ Πρόεδρε. με λίγο για την επιταχυμένη διαδικασία με την οποία έφτασε αυτό ενώπιον της Επιτροπής. Πολύ θα ήθελα να έχουμε αντίστοιχη αυροφροσύνη και σε άλλα μέλη όταν θέλουν να επιταχύνουν ε, τη διαδικασία τους. Δεν είχαμε καμία ε, δυνατότητα τροπολόγησης και συμπεριλαμβάνονται και κάποια στοιχεία που δεν ισχύουν. Ας πούμε ο έλεγχος ε, της ΕΠΑ από το Κοινοβούλιο, αν κοιτάξετε τις συνθήκες, θα διαπιστώσετε ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι συμβουλευτικός και ότι απλώς ενημερώνεται το Κοινοβούλιο και μπορεί να κάνει και ερωτήσεις. Μέχρι εκεί είναι η εξουσία στην ΚΕΠΑ και στην ΕΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχει καθόλου ρόλο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Όπως και πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός ε, σχετικά με τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου και ε, από πλευράς ορισμένων μελών. Αυτά ξεπερνούν ακόμα και τα όσα ορίζουν οι συνθήκες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταφ. Πρόεδρε. Ε, όντως, θεωρώ και εγώ ότι η διαδικασία ε, που ακολουθούμε είναι λίγο εκτός της πεπατημένης. Γεγονός όμως είναι ότι διεξάγεται ε, μία διαπραγμάτευση αυτό τον καιρό μεταξύ του Κοινοβουλίου μας και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και είναι σημαντικό εμείς ως Επιτροπή, αλλά και η Ολομέλεια, να ανταποκριθούμε, να απαντήσουμε στην πρόσφατη συνεδρία της ΚΟΖΑΚ και να προετοιμάσουμε το Κοινοβούλιο και για ε, τις απόπειρες της Πολωνικής Προεδρίας να ανταποκριθεί ε, στην υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη για να βελτιώσει τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Και θα ήθελα να πω στον Τζέφρι Βαν ότι το Κοινοβούλιο έχει ευρείες ε, δημοσιονομικές εξουσίες ε, και στην ΚΕΠΑ και στην ΕΠΑ στις αποστολές τους. Και θα ήταν για μας επιπόλαιο να τις παραβλέψουμε. Το πρωί συζητήθηκε το θέμα και η εντύπωση που αποκομίσαμε ήταν ότι το σχέδιο αντικατόπτριζε μια μεγάλη συνένεση στην Επιτροπή μας. Βεβαίως όποιος διαφωνεί μπορεί τώρα να το δηλώσει. Eh, Καλώς σημειώθηκαν οι απόψεις σας, είναι λογικότατες και αποδεχτές από διάφορες πλευρές σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής. Εμείς όμως είχαμε μια προθεσμία πάρα πολύ στενή εδώ σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας της Πολωνικής Προεδρίας. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα τεθεί σε ψηφοφορία τον μήνα Ιούλιο στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο και αυτή η διαδικασία λοιπόν επιτάχυνσης και με οι οποίες στην ουσία περιορίστηκαν εδώ, έχετε δίκιο. Σημερίζομαι λοιπόν πολλές από τις απόψεις σας ότι η πρακτική που ακολουθήσαμε δεν ήταν η κατάλληλη και ε, δεν θα πρέπει ίσως να επαναληφθεί όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι βέβαια Κανονικά θα έπρεπε να μπορούσαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να υπάρξει μεγαλύτερη προθεσμία για τις τροπολογίες, να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων. Επαναλαμβάνω, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή ήταν επιταχυμένη, αλλά ακριβώς για το λόγο τον οποίο ακούσατε, για να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία στην επερχόμενη Πολωνική Προεδρία. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία παρακαλώ. Θα υπάρξει μια ψηφοφορία συνολική θα έλεγα των διαφόρων παραγράφων. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στη διαδικασία αυτή, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν on block όλες τις τροπολογίες, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, ηλεκτρονική ψήφος τώρα για την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος συνάδελφος έβαλε την κάρτα του αλλά δεν ψήφισε ακόμα. Πέρα στις ψηφοφορίες. 44 ε, υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Έγινε δεκτό το ψήφισμα.